Thank you and welcome. Καλώς... Ε, Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία και κύριοι συμπρόεδροι, αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω σε αυτή την μήνυα κράση για το σεβασμό της δημοκρατίας των ολικών ελευθεριών του κράτους δικαίου, τρόλο της δικαιοσύνης. Και ευχαριστώ τους συγκεκριμένους ομιλητές μας που ήρθαν να μας μιλήσουν και να μας φωτίσουν με τις γνώσεις τους. Ευχαριστώ και την κυρία Χιουμπνέρ, την πρόεδρο της Επιτροπής, ε, που επέτρεψε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Επιτροπής Αύκο να γίνει αυτή η μήνυα ακρόαση. Και βέβαια όλους σας για την εξαίρετη συνεργασία. Ο κύριος Μωράης ε, σας ε, στέλνει τις, τη συγνώμη του καταρχάς που δεν μπορεί να είναι εδώ. Θα τον αντικαταστήσω εγώ άριθμα ψηφίσματα που έχει οθετήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναλημμένο ζητούν η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσει αποτελεσματικού μηχανισμού σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να παρακολουθείται σε μόνιμη βάση η τήρηση από τα κράτη-μέλη των θεμελιωδών αξιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω αυτέ έχουν καταγραφεί στο άρθρο 2 τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφεύγοντας ε, διπλά μέτρα και σταθμά και εξασφαλίζοντα μέσω ενό ε, συστήματο έγκαιρη προειδοποίηση, ε, το σεβασμό τη Δημοκρατία, κράτου δικαίου και θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Μάρτιο του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια ανακοίνωση για ένα νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν συστημικοί κίνδυνοι για, ε, που θα απειλούσαν το κράτος δικαίου, αναλαμβάνοντας έτσι διάλογο με τα κράτη-μέλη που είχαν ε, κινητοποιηθεί σε σχέση με τις εξελίξεις της προσφατές στην Πολωνία. Το Συμβούλιο λοιπόν ήδη είχε κάνει ένα πρώτο γύρο ε, σχετικό με το κράτος δικαίου υπό την Λουξεμβουριανή Προεδρία. Συνεχίζει τώρα με την Ολλανδική Προεδρία και με δεδομένο αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέθεσε το προηγούμενο Ιούνιο στην Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών να συμβάλλει και εκείνη στην ανάπτυξη και την ε, κατάρτιση ενό μηχανισμού, την επεξεργασία ενό μηχανισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Δημοκρατία, το κράτο δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα με τη μορφή μια νομοθετική έκθεση ίδια πρωτοβουλία. Έτσι λοιπόν, ξεκινούμε με το άρθρο 225 ε, τη Συνθήκη τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την έκθεση ίδια πρωτοβουλία, με τα 8 έγγραφα εργασία που παρουσιάστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών που ε, έχουν καταρτιστεί από, τον, ε, από την συγκήτρια από τους και και την συγκίτρια από την Επιτροπή ΑΦΚΟ για μια γνωμοδότηση που θα εξετάσει διάφορα θέματα για ένα μελλοντικό πλαίσιο σχετικό με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα που θα περιλαμβάνει το, ε, που θα καλύπτει μάλλον το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης, φασταμένους μηχανισμούς ευρωπαϊκού και διεθνούς επίπεδου, το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων, καθώς και τον ρόλο των δικαστηρίων και τις προκλήσεις που αυτά αντιμετωπίζουν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, Χρειάζεται βέβαια να εξηγήσω πόσο σημαντικό είναι ο ρόλο τη δικαστική εξουσία, πόσο μεγάλε είναι οι προκλήσει σε εθνικό επίπεδο, με βάση βέβαια και ανάλογα με την κάθε εθνική παράδοση. Οι διαφορετικοί μηχανισμοί στοχεύουν στην εξασφάλιση των αρχών τη διάκριση των εξουσιών, την ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη και την απόδοση δικαιοσύνης. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Χιούμπνερ για να συνεχίσει. Θα ήθελα και εγώ να πω εξ ονόματος της ε, ΑΦΚΟ ότι είμαστε ιδιαίτερω ευτυχείς ε, που συνεργαζόμαστε μαζί σας. Είναι μια πάρα πολύ καλή συνεργασία ε, και οπωσδήποτε επικοδομητική και ελπίζουμε καρποφόρα. Εμείς και από πλευράς της ΑΦΚΟ συμφωνήσαμε με τον Κλοντ Μωράες έτσι ώστε να έχουμε γενικά πιο στενή και πιο σε βάθος συνεργασία και όσον αφορά την γνωμοδότηση του ε, George Sheffling και νομίζω ότι αυτό ενισχύει την, τον διάλογο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρέπει να σας πω ότι και ο George Sheffling στην προηγούμενη συνεδρίαση της ε, ε, κοινοβουλευτικής μας επιτροπής παρουσίασε το έγγραφο αυτό σχετικά με μια πανευρωπαϊκή συζήτηση και διαδικασία και διάλογο πανευρωπαϊκή κοινοβουλευτική συζήτηση ε, και ε, επομένως ε, είναι πολύ σημαντικό που τώρα φτάνουμε σε αυτήν την ακρόαση. Φαντάζομαι ότι όλοι συμφωνείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση δικαίου σαφώς προορισμένη να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Βεβαίως έχει και το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά πέραν αυτού τα κράτη-μέλη έχουν μακρά δικαϊκή ε, παράδοση ε, φαντάζομαι ότι γνωρίζετε ότι τα ε, κράτη-μέλη όταν γίνονται μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πρέπει οπωσδήποτε να δηλώσουν σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Ο σεβασμός βεβαίως των θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει θεμητά να επιβάλλεται και στα κράτη-μέλη Υπάρχουν κάποια άρθρα στις ε, ε, συνθήκες που είναι ιδιαιτέρως ε, βαριά και σημαντικά και επομένως θα πρέπει να τα προσέξουμε. Το, η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο έχουν σκεφτεί τους επιπλέον μηχανισμούς μέσω των οποίων μελλοντικά προβλήματα θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν ε, καλύτερα και ε, βεβαίως να μην ε, υπάρχει κανένα κενό στα πλαίσια των πολιτικών και λοιπόν αλλαγών στις χώρες μέλη και ότι είμαστε βέβαιοι ότι πάντα θα διασφαλίζονται και θα είναι εγγυημένα τα θεμελιώδη δικαιώματα και ότι βεβαίως και η νομοθετική ε, και η εκτελεστική εξουσία ε, θα έχουν ε, μια κοινή βάση όσον αφορά την εγγύηση και την προστασία αυτών των δικαιωμάτων. Αυτά ήθελα να σας πω, δύο λόγια λοιπόν για το θέμα αυτό και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τη διάρκεια των εισαγωγικών παρατηρήσεων ε, να πω ότι έχουμε προσώπους ε, από όλες τις πολιτικές ε, ομάδες και επομένως είμαστε εδώ όλοι περιμένοντας να ακούσουμε τους ομιλητές μας έχουμε προσώπους από ευρωπαϊκά δικαστήρια, από εθνικά δικαστήρια, έχουμε δικαστές από ανώτατα δικαστήρια. Θα ήθελα αμέσως να δώσω το λόγο στην Αγγέλικα Νούσμπερκ, δικαστή από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ε, πρέπει να πω ότι ε, μετά το τέλος ε, της παρέμβασής της θα κάνουμε μία μικρή, θα δεχθεί ορισμένες ερωτήσεις έτσι ώστε να μπορέσει να απαντήσει ερωτήσεις που είναι μόνο για αυτήν. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ που μου επιτρέπετε να πάρω πρώτη το λόγο γιατί πρέπει να επιστρέψω στο Στρασβούργο έγκαιρα σήμερα για να είμαι και αύριο το πρωί. Πολύ χαίρομαι λοιπόν που έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαίρομαι που μπορώ να σας μεταφέρω κάποιες ιδέες από το Στρασβούργο. Δεν χρειάζεται βέβαια να φέρουμε γλάφκα εις Αθήνας εδώ, ούτε να επανεφεύρουμε τον τροχό. Θέλω να αναφέρω κάποια πράγματα, κάποιους προβληματισμούς. Πρώτα απ' όλα, σε τι βαθμό το δικαστήριο του Στρασβούργου έχει πετύχει μια ευρωπαϊκή συνένεση για το κράτος δικαίου. Και το δεύτερο, πώς η συνένεση αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να εκπονηθούν δίκτες και βάσει αυτό να προχωρήσουμε. Για την συνένεση όσον αφορά το κράτος δικαίου στην Ευρώπη πρώτα. Εδώ θέλω να τονίσω ότι για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το κράτος δικαίου είναι η βασική αρχή πάνω στην οποία βασίζεται κάθε άρθρο. Η σύμβαση αυτή βασίζεται στο κράτος δικαίου. Αυτό είναι το πνεύμα της. Τώρα βέβαια για να λειτουργήσουν όλα αυτά πρέπει να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία που έχουμε από την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων βάσει τεσσάρων ε, εγγύσεων και δύο θεσμικών εγγύσεων. Οι ουσιαστικές είναι η ισότητα, η βεβαιότητα, η ισότητα, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, το δικαίωμα σε δίκαια δίκη και η αναλογικότητα. Αυτές είναι οι ουσιώδεις, οι θεμελιώδεις εγγύσεις και επιτεθεσμικές είναι η ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος και η αποδοχή των αποφάσεων. Δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, οπότε επιτρέψτε μου να σας ε, δώσω τις κύριες γραμμές. Πρώτον, για την βεβαιότητα και την ομοιότητα. Είναι βασικές αρχές του κράτους και Πρέπει να γνωρίζουμε δηλαδή τι λέει ο νόμος και πώς αυτός εφαρμόζεται. Για το δικαστήριο όμως λοιπόν δεν ε, χρειάζεται μόνο ο νόμος αλλά και η ποιότητα του νόμου κάθε φορά που υπάρχει κάποια παραβίαση. Για παράδειγμα, ένα από τα προβλήματα του κράτους δικαίου είναι εάν οι έννοιες που περιλαμβάνονται στην ομοθεσία είναι κάπως ασαφείς. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα πολύ βασικό σε σχέση με το κράτος δικαίου και έχει να κάνει και με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Είναι το εξή. Πότε μπορείτε να διώξετε έναν δικαστή. Κυρίως στις χώρες μετά την Σοβιετική Ένωση υπάρχει η έννοια αυτή σε περίπτωση που υπάρξει παραβίαση του κράτους δικαίου. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ ευρύ, είναι πάρα πολύ γενικό σαν διατύπωση. Έχουμε λοιπόν νομολογία για την Ουκρανία. Υπήρξε εκεί πέρα μια περίπτωση τέτοια δικαστή, ο οποίος απολύθηκε επειδή παραβίασε την νομοθεσία και εδώ θα αναφέρω ένα κομμάτι μόνο της απόφασής μας για να σας δείξω ότι η νομική βεβαιότητα είναι κάτι αναγκαίο για το κράτος δικαίου. Λέει λοιπόν και παραθέτω. Η απουσία κάθε κατευθυντήριας γραμμής και πρακτική που έχει να κάνει με την περιορισμένη ερμηνεία της παραβίασης του όρκου και την ε, έλλειψη ρητρών ασφαλείας είναι πράγματα, πράγματα τα οποία οδηγούν σε απρόβλεπτες επιπτώσεις. Θα μπορούσαμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι κάθε κακή συμπεριφορά δικαστή η οποία λαμβάνει η χώρα οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του μπορεί να ερμηνευτεί, εάν το επιθυμεί το πειθαρχικό σώμα, σαν αρκετή βάση για πειθαρχικέ κυρώσεις που απορρέουν από παραβίαση του όρκου. Αν δηλαδή βλέπετε δεν υπάρχει συγκεκριμένη βάση για να απολύσετε έναν δικαστή, τότε η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης τίθεται υπό Νομική βεβαιότητα λοιπόν είναι κάτι αναγκαίο. Νομιμότητα και βεβαιότητα. Το δεύτερο είναι η ισότητα. Και εδώ θέλω να αναφερθώ στη χειρότερη πιθανότητα που είναι η εντελώς αυθαίρετη εφαρμογή της νομοθεσίας. Το δικαστήριό μας δεν εξετάζει την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας παρά μόνο εάν πρόκειται για αυθαίρετη εφαρμογή. Και εδώ έχουμε νομολογία πάνω σε αυτό και αυτή απορρέει από την Τσετσενία περίπτωση της Ρωσίας δηλαδή, όπου το δικαστήριο, και εδώ πάλι παραθέτω την ε, νομολογία του δικαστηριού μας, λέει ότι σύμφωνα με το δικαστήριό μας είναι εντυπωσιακό ο τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η νομοθεσία. Οι αποφάσει των ε, εσωτερικών δικαστηρίων μπορούν να κρυθούν ως αφαίρετες. Έχει να κάνει δηλαδή με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η νομοθεσία που είναι αυθαίρετος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο. Και υπάρχει και μια άλλη περίπτωση σπάνια στην ομολογία μας είναι όταν λέμε ότι ένα μέτρο χρησιμοποιείται με πολιτική διάθεση πολιτικοποιείται δηλαδή η απόφαση. Πρόκειται για το άρθρο 18 λοιπόν, το οποίο απαγορεύει να χρησιμοποιούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρόπο όχι ξεκάθαρο. Έχουμε εδώ την σαφή περίπτωση και γνωστή της αντιπολίτευσης στο Ασμπαϊτζάν, όπου εφαρμόστηκε το άρθρο 18 και οδήγησε στην κράτηση του κυριωμάτου. Αυτά λοιπόν είναι παραδείγματα για το η δεύτερη περίπτωση, το δεύτερο σημείο το οποίο σας ανέφερα που έχει να κάνει με την ισότητα σε αντίθεση με την αυθαιρεσία. Το τρίτο είναι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και το δικαίωμα σε δίκαια δίκη. Εδώ έχουμε μια αρκετά πλήρη νομολογία. Το άρθρο 6 αναφέρει ε, το δικαίωμα σε δίκαια δίκη και το τεκμήριο αθωότητας και έχουμε αναλύσει το κατώτερο επίπεδο εγγύησης. Αν γίνει έκδοση κάποιου, θα πρέπει να υπάρχει εγγύηση για δίκαια δίκη. Και το τελευταίο είναι η αναλογικότητα όπως σας είπα πριν. Και αυτό είναι κόκκινη γραμμή στην ομολογία του δικαστηρίου μας. Πάντα δηλαδή πρέπει να ζυγίζεις τα δικαιώματα του ατόμου και τα δικαιώματα της κοινότητας, της κοινωνίας και εκεί να βρεις την κατάλληλη λύση στο πρόβλημα. Ένα γνωστό παράδειγμα είναι εκείνο της Μπούρκα. Κατά πόσο δηλαδή ε, εμποδίζει την ε, συμβίωση σε μια κοινότητα ανθρώπων με και χωρίς. Αυτά λοιπόν είναι τα ουσιώδη. Και ερχόμαστε τώρα στα θεσμικά που είπαμε ότι είναι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης πρώτα απ' όλα. Το δικαστήριο για την δικαιοσύνη και τις θεμελιώδεις αρχές μέσα σε ένα κράτος δικαίου. Το πρώτο θέμα είναι λοιπόν η ύπαρξη μιας δικαιοσύνης η οποία έχει τη βούληση να δράσει σε περίπτωση που έχουμε παραβίαση δικαιωμάτων. Πρέπει να το κάνει, πρέπει να είναι αυτή η συνέπεια. Αν υπάρχει λοιπόν ένα έγκλημα πρέπει να υπάρξει η ανάκριση, οι δίκες διαδικασίες. Η ύπαρξη όμως της δικαιοσύνης αποτελεί τη βάση και μετά περνάμε στην ανεξαρτησία που έχει να κάνει με το πώς ορίζονται τα μέλη του δικαστικού σώματος, πώς ε, αντιμετωπίζουν και αντιστέκονται σε εξωτερικές πιέσεις. Το θέμα της ατιμορρησίας όποιος κρίνεται πρέπει να έχει την βεβαιότητα ότι οι δικαστές είναι ανεξάρτητοι. Αυτό ήταν το πρώτο θεσμικό ζήτημα. Και το δεύτερο είναι ότι το κράτος δέχεται έλεγχο απ' έξω. Δέχεται την ομολογία σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αποφάσεις του δικαστηρίου μας. Στα πλαίσια αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας ε, δώσω κάποια δείγματα για το πόσο μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει την πολυπλοκή αυτή νομολογία που διαθέτουμε εμείς στο Στρασβούργο. Όταν λοιπόν θέλετε να καθορίσετε τους δείκτες για σας, για τις δικές σας διαδικασίες, θα μπορούσατε για παράδειγμα, να δείτε τι παραβιάσεις έχουν εντοπιστεί. Και μπορείτε να το κάνετε αυτό είτε χώρα, να έχετε δηλαδή επισκόπηση αναχώρα και να δείτε τι παραβιάσεις βρίσκεται σε κάθε χώρα, αναχώρα, θα μπορούσατε επίσης να εξετάσετε όχι μόνο τις παραβιάσεις, αλλά και την συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις. Και εδώ είναι που εντοπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα βρίσκουμε πολλά προβλήματα στις χώρες μέλη, που μάλιστα είναι και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα έλεγα εδώ η προσέγγιση να είναι καθαρά στατιστική, δηλαδή να καθίσει κανείς να μετρήσει τις παραβιάσεις, δεν έχει και πολύ νόημα κάτι τέτοιο, γιατί αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, από τους δικηγόρους, πόσο καλή όχι είναι. Υπάρχουν θέλω να πω πάρα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν ένα στατιστικό αποτέλεσμα. Για μένα ο καλύτερος τρόπος είναι να δείτε τι είδους παραβιάσεις γίνονται. Είναι παραβιάσεις που έχουν να κάνουν με το πόσο κρατάει δίκη, κάτι το οποίο εντοπίζουμε περίπου σε όλες τις περιπτώσεις, που είναι ένα κακό φυσικά ε, σημάδι, αλλά δεν πρόκειται για πραγματικά παραβίαση της δίκης, ότι γίνεται δηλαδή μια δίκη που δεν είναι δίκαια, αλλά το ένα άλλο το άλλο. Μπορείτε επίσης να προσπαθήσετε να εντοπίσετε τι θέλετε να λάβετε υπόψη σας. Σε πολλές χώρες έχουμε προβλήματα με τις ηθίκες κράτησης. Άρα εδώ πέρα γίνεται παραβίαση όσον αφορά την, ε, τις συνθήκες κράτησης. Και κάτι χειρότερο, αν υπάρχει μεταχείριση... από τους ίδιους τους υπεύθυνου για την συμμόρφωση στον νόμο, αυτό είναι πιο σοβαρό. Οπότε πρέπει να δείτε τι παραβιάσεις ανακαλύπτεται στην κάθε χώρα και μετά να δείτε ποιες είναι οι πιο σοβαρές για να καταλάβετε σε τι βαθμό παραβιάζεται το κράτος δικαίου, γιατί αυτό είναι που θέλετε να αξιολογήσετε από ό,τι έχω καταλάβει. Μπορείτε επίσης να δείτε και το θέμα της συμμόρφωσης στις αποφάσεις τις δικαστικές. Είχαμε προβλήματα σε μια χώρα όπως είναι η Ρωσία που τώρα έχει ένα μηχανισμό για τις περιπτώσεις μη τήρησης, μη συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις. Το σταγματικό δικαστήριο μπορεί να κρίνει κατά πόσο έχει γίνει αυτό ή όχι. Είναι ο μοναδικός μηχανισμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν σημαίνει βέβαια ότι άλλες χώρες δεν θέλουν να εφαρμόζουν την ε, νομοθεσία μας τις αποφάσεις μας. Οπότε, για να παριθμίσουμε χώρες με προβλήματα όσον αφορά την ε, εφαρμογή μιας δικαστικής απόφασης είναι η Ιταλία, η Τουρκία, η Ρωσία, η Ουκρανία. Η Ιταλία είναι η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Βουλγαρία που είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς βρήκαμε ότι εκεί σε αυτές τις χώρες υπάρχουν συστημικά προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων. Όταν λοιπόν καθορίσετε τις διαδικασίες σας θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε και την εμπειρία που έχει το δικό μας δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων γιατί εμείς έχουμε συγκεντρώσει την ομολογία και έχουμε και στοιχεία και για τις 28 χώρες που σας ενδιαφέρουν εσάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτηση αυτή. Τώρα καλό τους συναδέλφους που θέλουν να διατυπώσουν ερωτήσεις προς την κυρία, προς την ε, δικαστή Σπέρκερ μόνο. Ο Γιολάινεν πρώτος και βέβαια καλό και τους λοιπούς συναδέλφους, εάν έχουν ερωτήσεις να σκάσουν το χέρι. Κύριος Λάιρεν, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Νοσπέρκερ, ευχαριστούμε πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα η τοποθέτησή σας. Είπατε πολύ σωστά ότι το κράτος δικαίου είναι βασική αξία στην οποία συνενούμε όλοι στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όσο και Ευρωπαϊκή Ένωση όλη στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο λοιπόν. Το θέμα είναι όταν παραβιάζονται οι αρχές του κράτους δικαίου. Πώς μπορούμε να το ελέγξουμε και πάνω απ' όλα τι με ποιο τρόπο μπορούμε να φέρουμε κυρώσεις. Και αυτό γιατί έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πρόβλημα. Οι μηχανισμοί που προβλέπονται από τις συνθήκες δεν επαρκούν για την επιτήρηση και μία σταθμισμένη επιβολή κυρώσεων, μια διαβαθμισμένη επιβολή κυρώσεων. Εσείς μας λέτε έχουμε τα πάντα στο Στρασβούργο, γιατί λοιπόν θέλετε και εσείς στις Βρυξέλλες να κάνετε το ίδιο πράγμα για δεύτερη φορά. Ναι. Ίσως αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μέλος, ήταν συμβαλόμενο μέρος στη σύμβαση, θα μπορούσαμε τότε με αίτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ζητήσουμε την ε, αντιμετώπιση μια υπόθεση παραβιασεων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κράτος δικαίου από κράτη-μέλη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ερώτηση ήταν αυτό. Ένα άλλο ζήτημα που προέκυψε πρόσφατα ήταν σχετικό με την ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη και την ελευθερία των μέσων μαζική ενημέρωση. Είναι δύο θέματα, θα έλεγα, πολύ σχετικά μεταξύ του, και εκτρώνουν κάνε όροι για την διαφύλαξη του κράτου δικαίου, όπω θεωρούμε εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε κάνει κάποιε συζητήσει για το πώ θα μπορούσε το, το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση παραβιάσεων των αρχών του κράτους δικαίου. Απάντηση. Θα είναι δύσκολο να σας μιλάω γιατί πρέπει να κοιτάω προς τα μπρος το μικρόφωνο ενώ βρίσκεστε πίσω μου. Θα μιλήσω γερμανικά πάντως για τα συγκεκριμένα προβλήματα, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης που αναφέρατε. Βλέπουμε νομίζω ξεκάθαρα τι μπορεί να κάνει το δικαστήριο και πώς μπορεί να σας υποστηρίξει και τι δεν μπορεί να κάνει. Μπορεί δηλαδή ατομικές προσφυγές να εκδικάσει με δεσμευτικό τρόπο έτσι έτσι ώστε τις ετοιμιγορίες του να τις αξιοποιήσετε και να καταλήξετε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα εσείς. Δεν μπορούμε όμως εμείς να κάνουμε αυτό που θα λέγαμε ένα screening, μια γενική επισκόπηση που συμβαίνει σε μια χώρα. Εμείς θα τη δούμε πάντα με μια ατομική προσφυγή που μας έχει υποβληθεί και έτσι θα μπορούσαμε τα αποτελέσματα αυτών των ε, εργασιών μας να τα εισάγουμε σε μηχανισμούς, σε έναν μηχανισμό. Αν και φαντάζομαι ότι αυτό σας ενδιαφέρει σας, γιατί έχετε και το άρθρο 7 του μηχανισμού που προβλέπει τον αποκλεισμό της συνθήκης, ε, αλλά δεν μπορεί ένα δικαστήριο ποτέ να κάνει μια γενική κρίση, να προβεί σε μια γενική κρίση. Μόνο με μονομένες περιπτώσεις μπορεί να κρίνει και με βάση αυτές να ορίσει προδιαγραφές που θα σας είναι χρήσιμες για το άρθρο 7. Και κατά τα άλλα ελπίζουμε πολύ σύντομα να γίνει μέλος και η Ευρωπαϊκή Ένωση της Σύμβασης. Ευχαριστώ κυρία Νετφέλτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ κυρία Νούσπερκερ για την παρουσίασή σας. Σύντομα κάποιες ερωτήσεις. Αναφερθήκατε σε κάποια βασικά στοιχεία, θεσμικές εγγύησεις πρώτα απ' όλα ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Και μας λέτε ότι είναι δυνατόν να αντληθούν κάποιες κοινέ προδιαγραφές σε σχέση με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης από την ομολογία του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου. Πολύ χρήσιμο αυτό γιατί είναι ε, κέριο ζήτημα. Όλα από εκεί ξεκινάνε και αν δούμε και τη συζήτηση που γίνεται με τον ορισμό νέου ε, δικαστή στον το Δικαστήριο Supreme Court στι Ηνωμένε Πολιτείε, ένα θέμα το οποίο έχει πολιτικοποιηθεί πολύ και κομματοποιηθεί σχεδόν ε, νομίζω ότι μπορεί κανείς να διερωτηθεί πολλά πράγματα. Εμείς έχουμε 28 χώρες μέλη με πολύ διαφορετικά συστήματα. Υπάρχουν όμως κάποια βασικά θεμελιώδη σημεία και στοιχεία. Δεύτερο, μας λέτε ότι δέχεστε αποφάσεις των κρατικών, των εθνικών δικαστηρίων. Με αυτό την αξιολόγηση αναχώρα. Όμως αυτό ε, δεν θα είναι ένα ζήτημα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όπου φαίνεται ότι το κοινο... η Επιτροπή και το Συμβούλιο μάλιστα ε, παραγνωρίζουν αποφάσεις ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και τις θεωρούν μάλλον φιλικές συστάσεις παρά δεσμευτικές δικαστικές αποφάσεις. Αυτή και μόνο η συμπεριφορά δεν υπονομεύει το κράτος δικαίου. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει το Δικαστήριο του Στρασβούργου για να βελτιώσει την τήρηση αυτών των αποφάσεων. Αυτό το πεδίο ακόμη δεν έχει διερευνηθεί. Και θα περιοριστώ σε αυτές τις δύο ερωτήσεις. Για την πρώτη σας ερώτηση, κοινέ προδιαγραφές, ανεξαρτησία του δικαστών. Ναι, βεβαίως, έχουμε αναπτύξει κοινέ προδιαγραφές. Η διαδικασία της απόλυσης, σε παραδείγματι, που έχουμε αντιμετωπίσει μερικές φορές απολύσεις και ξέρετε μέσω των πειθαρχικών επιτροπών ε, που έχουν προκύψει ε, έχουμε επισημάνει ότι πρέπει αυτές τις προδιαγραφές που θα οδηγήσουν σε απόλυση να τις ορίζουν οι ίδιες οι δικαστικές επιτροπές, οι πειθαρχικές επιτροπές για τους δικαστικούς και να μην υπαγορεύονται από την εκτελεστική εξουσία. Βεβαίως έχουμε πολλές φορές δει τέτοιου είδους μεμονωμένες περιπτώσεις. Έχουμε την υπόθεση υπάκαπης ε, κατά της Ουγγρικής ε, Δημοκρατίας. Ξέρετε ότι καταργήθηκε με την τροποποίηση του, της δικαιοσύνης το ανώτατο δικαστήριο, άρα έπαψε να υφίσταται. Και ω εκ τούτου απελήθη ο πρόεδρό του, ο οποίο προσέφυγε στο δικό μα δικαστήριο μιλώντα για παραβίαση τη ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη, δεδομένου ότι έχασε την εντολή του λόγω της αλλαγής ε, του συντάγματος της χώρας. Ε, εκκρεμεί αυτή η υπόθεση ακόμη, αλλά με αυτήν, και αυτό είναι και το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε, πρόκειται να περιγράψουμε και να προσδιορίσουμε τι συνέπειες μπορεί να έχει για το δικαστικό σώμα το ίδιο μια συνταγματική αναθεώρηση ή αλλαγές στο Σύνταγμα. Και βέβαια τι συνέπειε μπορεί να έχει για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Άρα ναι, προδιαγραφές έχουμε, είναι να εξελίξει όμω, είναι ρευστέ αυτέ οι προδιαγραφές ε, στην ομολογία μα. Για τη δεύτερη περίπτωση συμφωνώ απολύτω. Εάν οι αποφάσει του δικαστηρίου είναι δικαστικέ πρέπει ε, να, είναι δεσμευτικές, πρέπει να είναι δεσμευτικές σε διεθνέ επίπεδο. Άρα εάν δεν τη σέβεται μια αρχή, ε, ένα κράτο, βρίσκεται σε παράβαση διεθνούς δικαίου και ω εκ τούτου μπορεί να γίνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Ευρώπης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ είναι διπτά. Πρώτον, λέτε ή να μην τι δέχονται ή να μην τι εφαρμόζονται. Εάν δεν δέχονται τις αποφάσεις, μπορεί αυτό να οφείλεται, μάλλον όταν δεν εφαρμόζουν τις αποφάσεις, αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν έχουν τα χρήματα να αποζημίωση, αλλά το πρόβλημα κυρίω το πιο σοβαρό ε, είναι το να μην δέχονται τις αποφάσεις και εδώ έχουμε να κάνουμε μια ευθεία αφισβήτηση του δικαστηρίου και εδώ έχουμε να κάνουμε μηχανισμούς όπου προσπαθούμε να δείξουμε ότι η ε, συντριπτική πλειονότητα των ε, δικαστικών αποφάσεων εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη αν και υπάρχουν ανησυχητικά πολλές αποφάσεις που δεν εφαρμόζονται και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις για πιο αποτελεσματική διαδικασία υλοποίηση σε συνεργασία με τα εθνικά, κοινοβούλια, με τα εθνικά δικαστήρια, με τα εθνικά συστήματα εκτέλεσης των αποφάσεων. Και αυτό βέβαια πάντα θα είναι ένα ζήτημα εάν ε, καταρχήν δεν δέχονται τις δικαστικές αποφάσεις. Δηλαδή αν δεν παίζουν θα λέγαμε με τους όρους του παιχνιδιού της αποδοχής του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σούπλιν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ ε, κύριε Νιουσμπερκ που είσαστε σήμερα εδώ. Ε, μιλήσατε για νομική ε, ασφάλεια, ασφάλεια του δικαίου μάλλον και νομίζω ότι αυτή συμφωνούμε όλοι ότι είναι μια εκ των ουκάνευ συνθήκη αν θέλουμε να έχουμε και κοινωνική προβλεψιμότητα. Α, όμως ε, έχω την εντύπωση ότι το ζήτημα της ε, ε, βεβαιότητας δημιουργεί κάποια προβλήματα ερμηνείας. Κυρίως δε υπό το φως αυτού που είπατε ότι η νομολογία και τα πρότυπά της και οι προϋποθέσεις της εξελίσσονται αλλά αυτό όμως αντιτίθεται στην αρχή της ε, ασφάλειας του δικαίου. Πώς αντιμετωπίζετε λοιπόν αυτό το ζήτημα της ερμηνείας, επικαιροποιείται κάποια στοιχεία ε, με κάποιες αλλαγές ας πούμε στο καταστατικό έγινε λόγος ε, προηγουμένως ε, στην περίπτωση των Ηνωμένων ε, Πολιτειών αλλά ερωτώ από πού προέρχονται τα κριτήρια ποιος καθορίζει τα κριτήρια δεν είναι εύκολη ερώτηση το καταλαβαίνω αυτό δεύτερον αναφερθήκατε σε καταχρηστικές και αυθαίρετες αποφάσεις ποιος όμως καθορίζει το την αυθαιρεσία τρίτη ερώτηση ελαφρώς μονομερής αναφέρεστε στην ε, αναλογικότητα αναλογικότητα ανάμεσα στην κοινότητα είπατε και το άτομο τι εννοείται κοινότητα Αυτά είναι θεμελιώδη ερωτήματα. Ε, ναι, ξέρετε και εγώ έχω κάποια εμπειρία δικαίου. Ναι, φαίνεται, φαίνεται, λέει ε, η κυρία Νίσμπεργκερ η νομική βεβαιότητα και η αλλαγή ε, το, της νομολογίας ε, είναι στοιχεία που αντιτίθενται κατά κάποιο τρόπο, είναι αντιφατικά μεταξύ τους. Ε, εμείς θεωρούμε ότι κυρίως στο ποινικό δίκαιο είναι σημαντικό να έχουμε μια συγκεκριμένη προσέγγιση. Η βασική προσέγγιση λοιπόν είναι ότι ε, ο κατηγορούμενος για ε, εγκληματική πράξη, για ποινικά κολάσιμη πράξη ε, είναι αυτός επί του οποίου θα πρέπει να εφαρμοστεί το άρθρο 7 της συνθήκης μας με αρκετά αυστηρό τρόπο. Το άλλο θέμα είναι ότι η φιλοσοφία του δικαστηρίου είναι ότι το δικαστήριο είναι ένα ζωντανό όργανο ε, και επομένως ε, μπορεί να αλλάξει κάποιες αρχές. Ε, στη δεκαετία του 90 ας πούμε υπήρχαν κάποια στοιχεία τα οποία δεν ήταν, μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά από την κοινωνία και που τώρα η κοινωνία τα δέχεται. Πάντα λοιπόν λέμε ότι θα πρέπει να παραμένουμε εντός των ορίων που έχουμε ήδη προαποφασίσει και θα πρέπει να δούμε όταν ε, ε, υπάρχουν ε, αντίθετες απόψεις με ποιο τρόπο θα γίνει η ερμηνεία του δικαίου και μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε στην ερμηνεία του δικαίου. Και επομένως να υπάρξουν κάποιες προσαρμογές, εάν και εφόσον αυτές είναι απαραίτητες. Όσον αφορά τώρα την αυθαιρεσία ναι, εμείς ε, χρησιμοποιούμε το στοιχείο αυτό ε, σε ακραίες περιπτώσεις, δεν είναι πολύ συχνό. Ε, όμως, εάν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο γραπτό δίκαιο, τον νόμο και την δυνατότητα ερμηνείας του νόμου, αν υπάρχει μεγάλη, μεγάλο χάσμα, τότε θεωρούμε ότι υπάρχει ευθερεσία στην απόφαση. Επίσης, εμείς βλέπουμε τους νόμους σε σχέση με την εθνική κοινότητα. Ε, ας πούμε, θα πρέπει σε μια περίπτωση γαλλική, θα πρέπει να δούμε ε, το γαλλικό νόμο και την γαλλική ε, κοινωνία και επομένως θα πρέπει να δούμε την αναλογικότητα ανάμεσα στο κομμάτι που αφορά τον νόμο γενικά και την κοινωνία και το άτομο το συγκεκριμένο. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε άλλη μία ερώτηση, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει ε, να λήξει η συζήτηση αυτή, έτσι ώστε να προχωρήσουμε. Παρακαλώ, κύριο κύριος Σόλτς. Μία ερώτηση για βασικό θέμα. Ε, αναφερθήκαμε και στη σχέση με το ΔΕ. Ποια είναι η σχέση μεταξύ των, ποια πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι η σχέση και ο ρόλος που θα πρέπει να παίξουν τα δύο δικαστήρια όταν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Χάρτα. Ποια είναι η αίσθησή σας. Ευελπιστώ ότι θα είναι... Ε, α, εννοείται μετά την... Ε, ε εννοείται μετά την προσχώρηση. η δικιά μας, ε, το δικό μας δικαστήριο ερμηνεύει την ε, ε, συνθήκη. Εμείς ερμηνεύουμε απλά την συνθήκη. Προσχώρηση σημαίνει ότι η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου μπορεί να αξιολογηθεί και επί τη βάση της συνθήκης. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Επομένως, κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει ε, δεν υπάρχει ασάφεια όσον αφορά τις κατεμέ σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες των δικαστηρίων και πιστεύω ότι η προσχώρηση αν συμβεί ε, θα ε, σημαίνει ότι τα πράγματα θα γίνονται ακόμα καλύτερα και θα λαμβάνουν χώρα με ακόμα πιο απλό τρόπο από ό,τι τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ λέει ο ευχαριστούμε πολύ για την συμβολή σας στην συζήτηση. Θα προχωρήσουμε τώρα, θα δώσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή, ο, πρόκειται για τον Γενικό Εισαγγελέα Μίκαλ Μπομπέκ, ε, του, ε, από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και μετά το, έχετε το λόγο κύριε Μπόμπεκ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε να μιλήσω σήμερα εδώ για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα το οποίο πραγματικά είναι άξιο συζήτησης και ιδιαίτερης προσοχής διότι αποτελεί την βάση για οτιδήποτε άλλο. Πριν ξεκινήσω θα ήθελα να σας δώσω κάποια ε, στοιχεία. Εγώ ε, ε βεβαίως ε, είμαι απεσταλμένος κατά κάποιο τρόπο από το δικαστήριο αλλά εδώ θα μιλήσω εξ ονόματός μου και επομένως θα αφήσω παραδίπλα την, τη θέση που έχω στο δικαστήριο. Μπορώ να απαντήσω βεβαίως και για θέματα τα οποία αφορούν εκκρεμείς υποθέσεις. Ε, επί της ουσίας τώρα. Έχω λίγο χρόνο στη διάθεσή μου και γι' αυτό αποφάσισα να ασχοληθώ με τρία ε, κεντρικά κατά την άποψή μου ζητήματα. Πρώτον, ε, θα κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις ε, σχετικά με το ιδιαίτερα υποβοηθητικό έγγραφο το οποίο μου αποστήλατε. Θα αν θέλετε να το σχολιάσω, μπορώ να το σχολιάσω. Δεύτερον, από τη στιγμή που η ακρόαση αφορά το ρόλο της δικαιοσύνης, ε, στα επόμενα σημεία μου θα ήθελα να ασχοληθώ ακριβώς με την δικαιοσύνη. Ε, ε, κυρίως όσον αφορά το δικαστήριο και το ρόλο που μπορεί να παίξει και τρίτον τη σχέση του με τα εθνικά δικαστήρια. Και βεβαίω, αν θέλετε κάποιες ερωτήσεις ή αν θέλετε να εστιάσω περισσότερο σε κάποια από στοιχεία που θα έχω αναφέρει, βεβαίω θα το κάνω. Τρει ε, παρατηρήσεις έχω όσον αφορά το έγγραφο εργασία ε, ε, για την ακρόαση, το οποίο θεώρησα πολύ σημαντικό. Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου ε, να πω ε, κάτι το οποίο σας περιμένετε να πει ένας ενιαρός δικηγόρος. Ε, η νομική βάση και η αρχή της νομιμότητας είναι πάρα πολύ σημαντική και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητώ συγγνώμη που το τονίζω γιατί υπάρχουν δύο δυνατότητες τροποποίησης των, των συνθήκων και επομένως θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να πούμε ότι η αρχή της νομιμότητας ισχύει και για, τις ευρωπαϊκές, και για τους ευρωπαϊκούς ε, θεσμούς. Αν θέλουμε να αναπτύξουμε κάτι ε, ε, καινούριο θα πρέπει οπωσδήποτε να μην ξεπεράσουμε τα εσκαμμένα και τις αρμοδιότητες. Δεύτερον όσον αφορά αυτό το έγγραφο είναι μια απλή ερώτηση ενδεχομένως πριν δημιουργηθούν νέες αρμοδιότητες και νέα πλαίσια, μήπως θα έπρεπε να δούμε με καινούρια ματιά ε, τα υφιστάμενα και να δούμε πώς μπορούν περαιτέρω να χρησιμοποιηθούν ε, στο έγγραφο ε, 7 αναφέρονται οι φυστάμενοι μηχανισμοί. Ε, ε, πολλά πράγματα αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο που ε, κανείς μπορεί να χρησιμοποιήσει εάν έχει τη διάθεση να το κάνει. Εγώ δεν νομίζω ότι μια απλή διαδικασία επί είναι κακό, κακή δυνατότητα εάν κανείς τη δει προσεκτικά. σε γενικές γραμμές οι διαδικασίες ε, επί παραβάση δίνει δυνατότητες και από τις δύο πλευρές. Ε, τα προηγούμενα χρόνια και αν δούμε τις ε, δημοσιοποιημένες πληροφορίες ίσως δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πλήρως Εάν δούμε τώρα τα αριθμητικά στοιχεία, βλέπουμε ότι οι διαδικασίες ε, επί ε, παραβάση ε, μειώνονται ενώπιον του δικαστηρίου, ενδεχομένως γιατί ο μηχανισμός βάσει της νέας συνθήκης Λισαβόνας είναι πιο αποτελεσματικός, αλλά μπορεί να ευθύνεται και σε κάτι άλλο ότι ενδεχομένως οι πίνακες αντιστοιχειών δεν είναι τόσο σαφείς ή είναι πολύ σαφείς ή οτιδήποτε άλλο και ε, φυσικά θα πρέπει ε, να δούμε εάν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να λειτουργήσουν να χρησιμοποιήσουμε τα, τα υφιστάμενα εργαλεία και να τα ε, λειτουργήσουμε καλά πριν δημιουργήσουμε καινούργια. Αλλά αυτό το βάζω σαν γενική ιδέα και από την άλλη πλευρά όταν ε, δεν υπάρχει ε, εισαγγελία ε, τότε μπορεί κάποια, κάποιες δύσκολες περιπτώσεις να μην προωθούνται γιατί κανείς δεν θα πάρει απόφαση από αυτόν. Και κάτι άλλο τώρα και βεβαίως χαίρομαι που έχω εδώ συναδέλφους από το Στρασβούργο ενδεχομένως σε βάθος συνεργασία, περισσότερη συνεργασία με το δικαστήριο του Στρασβούργου θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε καλύτερη συνεργασία ίσως όχι όσον αφορά το προήμιο και τις αιτιολογικές σκέψεις, αλλά όσον αφορά το κυρίως σώμα. Ακούσαμε ενδιαφέροντα πράγματα για το κεκτημένο του Στρασβούργου. Υπάρχει βέβαια ε, και πολύ συγκεκριμένη εντολή όσον αφορά τα ζητήματα αυτά ε, και νομίζω ότι μπορεί να προστρέχουμε σε αυτήν ε, πιο συχνά. Το κάναμε το 2004 είχαμε καλή συνεργασία όσον αφορά τις προενταξιακές συνθήκες κλπ. Αυτές ήταν μερικές σύντομες παρατηρήσεις όσον αφορά το ε, ενδιαφέρον έγγραφο το οποίο μου στείλατε. Δεύτερον, μια και μιλάμε για δικαστήρια, να πούμε τι μπορούν να κάνουν τα δικαστήρια αυτά η ενδυνάμει συμβολή ε, ε, ε, περιορίζεται λόγω συγκεκριμένων αρχών και περιορισμών. πρώτα απ' όλα και συγγνώμη που είμαι κοινότοπο, πρέπει να υπάρχει υπόθεση. Δεύτερον, θα πρέπει να είναι αρμόδια για την υπόθεση το δικαστήριο. Από αυτή την άποψη, οι, οι ίδιες οι αρχές οι οποίες περιορίζουν εσά περιορίζουν και το δικαστήριο, το Συμβούλιο, η Κομισιόν. Ε, αυτό βεβαίως ε, δεν μπορεί να ε, εμποδίσει κάποιες υποθέσεις οι οποίες είναι ιδιαίτερως προβληματικές, οι οποίες αφορούν παραβίαση δικαιωμάτων ή παραβίαση του κράτους δικαίου από πλευρά των κρατών, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι τα πράγματα δεν είναι, είναι πολύ σαφή όσον αφορά. Όσον αφορά τώρα το επίπεδο του δικαστηρίου, δεν πρέπει να υποτιμώνται οι τεχνικές υποθέσεις και ε, στο ενδιαφέρον έγγραφο ε, παρατήρησα μία ελαφρά ε, υποτίμηση αυτών των τεχνικών υποθέσεων. Βεβαίως εξαρτάται από το τι προσέγγιση παίρνει ο καθένας. Μερικοί θέλουν πολύ μεγάλα βήματα, ενώ άλλοι θεωρούν ότι μέσω μεμονωμένων υποθέσεων, έστω που αντιμετωπίζουν πιο τεχνικά ζητήματα, μπορεί κανείς να προχωρήσει. Παράδειγμα, Ε, συζητήθηκαν ας πούμε περιπτώσεις όπως ε, ε, Κομισιόν ε, κατά Ουγγαρίας ε, επίσης το θέμα των, της επιμήκυσης ε, της ε, συνταξιοδότησης επί δεκαετία θέματα τα οποία είναι, μπορεί να είναι τεχνικά αλλά τα οποία βασίζονται σε, σε ανεξαρτησία των προσωπικών δεδομένων περίπτω υπόθεση Κομισιόν Αυστρία, Κομισιόν Ουγγαρία ε, και ε, εξού και το ερώτημα ε, πρέπει να προχωράμε μέσα από τέτοιου είδους βαριές δραματικές περιπτώσεις βάσει του άρθρου 2 ας πούμε μπορεί να υπάρχουν και άλλες παρόμοιες υποθέσεις παραδείγματα που προέρχονται από τα εθνικά δικαστήρια. Άλλο παράδειγμα το άσυλο δικαίωμα ασύλου αιτήματος ασύλου διοικητικά ζητήματα περιορισμοί αμοιβαίας αναγνώρισης ε, για βάση κάποιων ε, παραβάσεων που έχουν διαπιστωθεί στις εθνικές διαδικασίες. Και έρχομαι στο δεύτερο ε, θέμα πολλά μπορούν να γίνουν ήδη βάση και εντός του υπάρχοντος συστήματος. Αν ξεσκονίσουμε λίγο τις δυνατότητες. Τρίτο και τελικό σημείο της ε, σύντομης παρουσίασής μου. Ποιος είναι ο ρόλος των εθνικών δικαστηρίων ή τι μπορεί να γίνει για τα εθνικά δικαστήρια από πλευράς ευρωπαϊκής. Και εδώ το σημείο αυτό δεν στο σημείο αυτό δεν μπορεί να αποδοθεί ε, υπερβολική σημασία γιατί υπάρχουν πρωτοβάθμια εθνικά δικαστήρια ε, όπου, ε, ε, όπου κατατίθενται όλα τα νομικά όπλα και οι νομικές διαδικασίες σε πρωτοβάθμιο επίπεδο και πρέπει να πω ότι κατά αυτή την έννοια θα πρέπει να αποδοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό το εθνικό πρώτο επίπεδο. Ε, εγώ προέρχομαι από το τσέχικο δικαστικό σύστημα και έχω κάποια εμπειρία όσον αφορά τα θέματα αυτά. Έχω και κάποια άποψη όσον αφορά τις ε, ε, μεταρρυθμίσεις του δικαστικού συστήματος στις νέες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κεντρική Ανατολική Ευρώπη. Στο έγγραφο που μου στείλετε αλλά και σε άλλα προηγούμενα έγγραφα της Κομισιόν πρέπει να πω ότι ε, αναφέρονται πολλά στοιχεία όπως scoreboard, πίνακας ε, επιδόσεων, ε, έλεγχος, εποπτεία, επιτήρηση κτλ. Εγώ όμως και για να διευρύνουμε λίγο τη σκέψη μας επί του θέματος θα ήθελα να σταματήσουμε να έχουμε μόνο αρνητικά στοιχεία. Ίσως να δώσουμε μια θετικότερη προσέγγιση και μία ε, θετικότερη έτσι όθηση ε, και πιστεύουμε ότι ίσως δεν θα πρέπει μόνο αναδρομικά ε, να κολλάμε σε αρνητικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να τιμωρηθούν αλλά να στραφούμε προς το μέλλον πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε νέες ικανότητες στο μέλλον ενδεχομένως αυτά που λέω να μην λύσουν τα παρόντα ζητήματα και την παρούσα κρίση. Ναι, αλλά εγώ προσπαθώ ε, να ε, στραφώ ε, προς το μέλλον και να δω με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε ενδεχομένως να αποφύγουμε νέες κρίσεις και αυτό μπορεί να γίνει μέσω οικοδόμησης ικανοτήτων στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να κάνω και κάποιες ε, γενικότερες ε, σκέψεις ε, και όχι μόνο προερχόμενος από νέα χώρα λέω ότι όντως μπορούμε να διαπιστώσουμε προβλήματα όσον αφορά την λειτουργία της δικαιοσύνης. Εγώ δεν λέω ότι κάθε κυβέρνηση θα λύσει οπωσδήποτε τα ζητήματα αλλά λέω ότι θα πρέπει να παρασχεθεί η απαραίτητη βοήθεια έτσι ώστε ε, να λυθούν, ε, να ενθαρρυνθεί ας πούμε η επιλογή των δικαστών ε, βάσει ελεύθερων διαδικασιών, ανεξάρτητων διαδικασιών, βάσει αξιοκρατίας. Δεύτερον, σε διαφορετικό επίπεδο ας πούμε, ίσως η δικαιοσύνη θα πρέπει να έχει δυνατότητα ας πούμε ε, συν ε, με την πολιτική διαδικασία δηλαδή ε, να δημιουργηθεί μια δομή δικαστική, δικαιική η οποία να βοηθάει και το κάθε ένα ε, άτομο. Ε, θα πρέπει να προχωρήσουμε με το λεγόμενο σύστημα checks and balances, ε, να δούμε κυρίως σε ορισμένα δυστυχώς νέα μέλη βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ ισχυρά δικαστικά συμβούλια τα οποία δεν ξεκουνιούνται με τίποτα. Τέλος, θα μπορούσαμε να ενθαρρύνουμε την δημιουργία δικτύων, ανταλλαγή γνώσης, όχι μονάχα στο ανώτατο δικαστικό επίπεδο, όχι μόνο σε ανώτερο επίπεδο, αλλά και σε πιο χαμηλό επίπεδο. Ε, γιατί ε, αν κάποιος ε, δικαστής υφίσταται πίεση είναι πάρα πολύ σημαντικό να αισθάνεται ότι δεν είναι μόνος του, ότι έχει μία στήριξη. Ε, εάν ένας ε, δικαστής ε, πρέπει να υψώσει το ανάστημά του απέναντι σε μια κυβέρνηση και να πει κάτι που δεν ευχαριστεί την κυβέρνηση αυτή. Είναι πολύ πιο σημαντικό να αισθάνεται ότι δεν δίνει τον αγώνα αυτό σε ένα γαλαξία έτη φωτός μακριά από τους υπόλοιπους. Όχι, ότι είναι κοντά, κοντά του και άλλοι. τι μπορούμε να κάνουμε ε, όσον αφορά ε, τις ενδεχόμενες αλλαγές των συνθήκων, εγώ θα έλεγα ε, σε, μια τέτοια, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο να μην δούμε μονάχα τις πιο σοβαρές περιπτώσεις ή τις πιο ισχυρές κυρώσεις, αλλά να δούμε και σε πιο μικρή κλίμακα στοιχεία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην γενικότερη αντιμετώπιση ε, του προβλήματος να μην δούμε μόνο τις κυρώσεις, να δούμε και την ε, θετική πλευρά και την οικοδόμηση ε, ικανοτήτων. Ε, εν είδη συμπεράσματος θα πω κάτι εντό εισαγωγικών τώρα έχουμε ε, δημοκρατία, α βρούμε και μερικού δημοκράτε. Αυτό το είπε το 1920 ένα πρωθυπουργό τη Τσεχία, αλλά ε, είναι δραματικά επίκαιρο νομίζω. Σα ευχαριστώ πολύ. Με χαρά σα ακούσαμε και του δύο. Όλοι νομίζω. Α ακούσουμε τώρα τον Ζαν Πρώτο πρόεδρο του αναιρετικού του Βελγίου αλλά και επικεφαλής της Ένωσης των Νότων Δικαστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, για την τιμή που μου κάνετε, που μου επιτρέπετε να εκφραστώ εδώ, από το βήμα αυτό στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το χρόνο που έχω στη διάθεσή μου θα ήθελα να τον αξιοποιήσω για να αναλογιστώ μαζί σας κάποιους αντικειμενικούς δίκτας, νομικούς δικαστικούς δίκτας, ακριβής. του οποίων πιστεύω αισθάνεστε την ανάγκη εν ώψη της ανάγκης να υποπτευθούν ορισμένα κράτη, εν πάση περιπτώσει συγκρίσεως σε σχέση με τις βασικές αρχές του κράτους δικαίου που συζητήθηκε από, τις, από τους προλαλήσαντες και σε αυτό θα ήθελα να τοποθετηθώ. Πρέπει να συνεννοηθούμε τι εννοούμε όταν μιλούμε για κράτος δικαίου. Κράτος δικαίου σημαίνει ένα κράτος να εγγυάται μια σειρά από δικαιώματα στους ειδικούς του, ταυτόχρονα όμως αποσιωπάτε μια πολύ σημαντική, εξίσου σημαντική με την πρώτη ε, απόφαση, ε, τοποθέτηση αρχή, ότι δηλαδή το ίδιο το κράτος υποτάσσεται στους κανόνες που το ίδιο έχει παραγάγει. Ποιοι είναι αυτοί λοιπόν οι αντικειμενικοί δείκτες που θα μας επιτρέψουν να έχουμε ένα σύστημα που θα λειτουργεί με βάση τις αρχές του κράτους δικαίου. Και εδώ νομίζω έχουμε δύο πτυχές. Αφενός μεν μάλλον δύο κατηγορίες πτυχών. Πρώτον λοιπόν έχουμε το σύνολο που χρειάζεται να οικοδομηθεί για να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας και μια και γίνεται λόγο σε δικαστική εξουσία, πρέπει να διαρωτηθούμε τι σημαίνει δικαστική εξουσία και ποια είναι τα κριτήρια. Και να πει κανεί ότι η εξουσία λέγεται δικαστική και δεν είναι απλώ μια διοικητική αρχή του κράτου που στόχο έχει να ε, διεκπεραιώνει ε, διαφορέ μεταξύ των πολιτών. Είναι ανεξάρτητη η δικαστική εξουσία. Τι καθιστά τη δικαστική αυτή η εξουσία ανεξάρτητη και τι εργαλεία έχει θέση τη για να διασφαλίζει αυτή την ανεξαρτησία. Να μια πρώτη λοιπόν κατηγορία πτυχών που πρέπει να εξεταστούν. Μια δεύτερη κατηγορία πτυχών πρέπει να εξεταστεί είναι εάν αυτή η δικαστική εξουσία, μπορεί μια και μιλούμε για δημοκρατία, να είναι σε θέση να διαδραματίσει αυτό το ρόλο της αντισταθμιστικής εξουσίας και με τι εργαλεία μπορεί αυτή η δικαστική εξουσία εάν υποθέσουμε ότι υπάρχει, να διαδραματίσει αυτό το ρόλο της αντισταθμιστικής εξουσίας που είναι απαραίτητος στην θεωρία της διακρίσεως των εξουσιών όπως την έχει διδάξει σε όλους μας ο Μοντεσκιό. Πρώτη λοιπόν κατηγορία εργαλείων, τα εργαλεία της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας που είναι πολύ σημαντική αρχή, δεν αποτελεί προνόμιο για τους δικαστές που απαρτίζουν αυτήν την εξουσία. Είναι πάνω απ' όλα ε, μια αρχή και μια εγγύηση που αφορά την ευθύνη τους και καταγράφεται στο άρθρο 6.1 της Σύμβασης για τη διαφύλαξη των, θεμελιωδών δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών. Τι σημαίνει όμως και σε τι συνίσταται αυτή η ανεξαρτησία. Αποτελεί εγγύηση λοιπόν για τον υπήκο ενός κράτου, για το υποκείμενο του δικαίου, ότι η απόφαση που θα ληφθεί και που θα πλήξει την ε, ε, τιμή, την αξιοπρέπειά του, την ελευθερία, το πορτοφόλι του, δεν θα ληφθεί παρά μόνο η απόφαση αυτή με βάση τα πραγματικά περιστατικά της διαφοράς και τα ένομα χαρακτηριστικά που εφαρμόζονται σε αυτήν και μόνο πάνω σε αυτά θα στηριχθεί η απόφαση. Ο δικαστής λοιπόν με την απόφαση του είναι ανεξάρτητος εφόσον είναι ασφαλής και προστατευμένος από οποιαδήποτε πίεση. Είτε αυτή είναι πολιτική ή ιεραρχική ή ηλική φύσεως. Για να δούμε αυτές τις πτυχές λοιπόν. Πολιτικής φύσεως ανεξαρτησία, ο Γενικός Εγγελέας το ανέφερε, η πολιτική ανεξαρτησία πρέπει να εξασφαλίζεται. Δεν είναι ουρανοκατέβατη όμως, δεν αρκεί να τη διακηρύσουμε για να υλοποιείται. Χρειάζεται εργαλεία, το είπατε και εσείς, και ένα από τα εργαλεία αυτά είναι μια ειδική διαδικασία, ιδιάζουσα διαδικασία ορισμού υποψηφιότητων, επιλογής και προαγωγής δικαστικών λειτουργούν με βάση κριτήρια, λειτουργών με βάση κριτήρια αντικειμενικά ικανοτήτων και ανεξαρτήτως ιασδήποτε επιρροής από ομάδες πιέσεως ή κόμματα στο Βέλγιο, από το οποίο και εγώ προέρχομαι, οι δικαστές διορίζονται και προάγονται από τον Βασιλέα με σύσταση, με βάση σύσταση ανεξάρτητου σώματος του οποίου την ύπαρξη το, το Σύνταγμα το λεγόμενο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Η ανεξαρτησία λοιπόν αυτή είναι συνδεδεμένη με την ανεξαρτησία των διορισμών και προαγωγών των δικαστικών λειτουργών και αυτό αποτελεί τη βάση και την απόλυτη απαρχή της ανεξαρτησίας. Η δικαστική εξουσία, αν θέλουμε να διαδραματίσει αυτό το ρόλο της αντισταθμιστικής εξουσίας, ε, και να διδραματίσει πλήρως το ρόλο της στην ενίσχυση τη δημοκρατία, τη λειτουργία της δημοκρατίας, θα πρέπει να χαίρει και μίας υλική ανεξαρτησία. Σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Βέλγιο ε, διαφαίνεται ένα κίνημα η δικαστική εξουσία να έχει αυτονομία ως προς τη διαχείριση του υλικού ε, των υλικών μέσων που έχει θέση τη και εδώ και θα ήθελα ίσως ε, να επισημάνω μια ανησυχία για τη βελγική εμπειρία να είναι χρήσιμη στις ε, σκέψεις σας για το Βέλγιο ειδικά λοιπόν το 2014 είναι έτος το οποίο καταγράφει την απώλεια για το Υπουργείο Δικαιοσύνης κάθε αυτονομία σε σχέση με την πρόσληψη προσωπικού. Είχαμε, και χρησιμοποιώ παρατατικό χρόνο, νόμους οι οποίοι ισχύουν ακόμη, δεν, δεν, είναι όμως ε, πλέον, δεν εφαρμόζονται πλέον, δεν είναι σεβαστοί, που όριζαν για κάθε δικαιοδοτική αρχή τον αριθμό των δικαστών, των γραμματέων, του διοικητικού προσωπικού, νομικές δηλαδή εγγυήσει που εξασφαλίζουν τον ρόλο, τον αριθμό των δικαστών, δικαστικών λειτουργών, τους οποίους τους κανόνες όμως δεν εφαρμόζει πλέον και δεν σέβεται το Βέλγιο παρότι παραμένουν ενισχύ οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις σε μια χώρα όπως η δική μου η οποία είναι υποτίθεται κράτος, δημοκρατικό κράτος δικαίου διαπιστώνεται πως ενδέχεται να υπάρξουν εξελίξεις οι οποίες μας προβληματίζουν σε σχέση με την υλική ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Άλλες ανησυχίες επίσης εκφράζονται σε σχέση με την αρχή της του αμετακίνητου των δικαστών. Δεν μπορεί να μετακινείται δηλαδή να ε, αποστέλλεται στη, σε κάθε γωνία του ορίζοντα ε, ένας δικαστής όπως οπωσδήποτε άλλος ε, δημόσιος υπάλληλο με μεταθέσεις. Δεν επιτρέπεται αυτό γιατί η εγγύηση για την ανεξαρτησία του δικαστή συνίσταται και στο ότι έχει το αμετακίνητο, δηλαδή μόνο με δική του συνένεση μπορεί να μετατεθεί. Αυτό είναι κανόνες που ισχύουν εδώ και 100 ε, και χρόνια και είναι σημεία ε, ισχυρά των εξελίξεων και πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη. Άλλο ανησυχητικό στοιχείο, το οποίο όμως ε, πιστεύω δεν είναι εύκολο να αναλυθεί εδώ λόγω χρόνου, είναι το ότι περνάμε από την χρηματοδότηση με βάση το κόστος ε, της λειτουργίας της δικαιοσύνης σε ένα σύστημα χρηματοδότησης με κλειστούς φραγισμένους φακέλους, πράγμα το οποίο μπορεί να επηρεάσει ασφαλώς την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Επίσης, σε ιεραρχικό επίπεδο, ε, ο ρόλος του δικαστή, η λειτουργία του δικαστή, ο, ο τρόπος του εκδικάζει, ε, η υπηρεσία, το, το λειτουργήμα του δικαστή δεν μπορεί να επάγεται σε ιεραρχικές κατευθύνσεις και δομές. Σε αυτό είμαστε πολύ επιφυλακτικοί εμείς στο Βέλγιο. Ένας υπουργός δηλαδή δικαιοσύνης ο οποίος αποτολμά να διατυπώνει επιφυλάξεις ή σχόλια σε, για δικαστική απόφαση η οποία ακόμη δεν έχει πάρει τη μορφή του δεδικασμένου θα ε, βρεθεί απολογούμενος από τη δικαιοσύνη θα κληθεί να δώσει δηλαδή εξηγήσει στους δικαστές. Δεν υπάρχει περίπτωση η εκτελεστική εξουσία να σχολιάσει εν εξελίξη ε, απόφαση, δίκη μάλλον. Για δε τις εισαγγελικές αρχές, για την δικαιοσύνη της έδρας, ε, υπάρχει διαφορετική κατάσταση στο Βέλγιο. Μπορεί να δώσει κάποιε συστάσεις ο Υπουργό Δικαιοσύνη, αλλά μόνο θετικέ, μόνο να οφείσει σε μία πράξη την εισαγγελική αρχή δεν μπορεί να απαγορεύσει στην εισαγγελική αρχή να αναλάβει μία δράση, μία πρωτοβουλία. Και βεβαίω η ανεξαρτησία ε, των, δικαστικών λειτουργών εκφράζεται και με άλλε αρχέ. Επί παραδείγματι, στο πειθαρχικό δίκαιο άκουσα μια τοποθέτηση νωρίτερα αλλά δεν ε, φαντάζομαι ότι μεταφράστηκε σωστά γιατί ακούστηκε η λέξη απόλυση δικαστή. Μα δεν είναι δυνατόν να απολυθεί δικαστή. Δεν μπορεί λοιπόν να απολυθεί ο δικαστής, να παυθεί μπορεί, απαγορεύεται να απολυθεί. Μπορεί λοιπόν να γίνει δίωξη πειθαρχική από έναν άλλο δικαστή όμως. Στο Βέλγιο έχουμε πειθαρχικά όργανα, δικαστικά πειθαρχικά όργανα, αρμόδια να απαγγείλουν πειθαρχικέ ε, κυρώσει ει βάρο ε, κατά των δικαστών, οι οποίοι έχουν σε θέσή το δικαίωμα τη προσφυγή κατά αυτών των αποφάσεων. Ένα δικαστή, σε παραδείγματι, θεωρήσει, εκτιμήσει ότι το μέτρο της, ε, των κατηθυκόντων που του ανατίθενται, τον ε, υποβιβάζει τρόπον την δηλαδή τοποθετείται σε ένα δικαστήριο, τμήμα δικαστηρίου ε, το οποίο θεωρεί ότι δεν τον ικανοποιεί και εφόσον είναι σε θέση να αποδείξει ότι αυτή η υποτιμητική τοποθέτηση συνιστά πειθαρχική και καλυμμένη πειθαρχική κύρωση έχει στη διάθεσή του προσφυγή, δυνατότητα προσφυγής ενώπιον του πειθαρχικού οργάνου. Πρώτη πτυχή λοιπόν η ανεξαρτησία πολιτική, ηλική, πειθαρχική, ιεραρχική ανεξαρτησία. Δεύτερη κατηγορία πτυχών, ο δικαστής, άπαξ και υπάρχει και υφίσταται η δικαστική εξουσία, πρέπει να της ε, ρόλος στην προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ζήτημα επίκαιρο λόγω και της τρομοκρατικής απειλής ε, ε, με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η δημοκρατία μας, οι δημοκρατίες μας. Τι εργαλεία λοιπόν για προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών έχει στα χέρια του ο δικαστής, μα κύριο εργαλείο για την προστασία αυτή είναι πιστεύω ο δικαιοδοτικός έλεγχος της συμβατότητας των διατάξεων των ε, ε, κανόνων του δικαίου με τους ιεραρχικά ανώτερους κανόνες. Αυτή είναι μια βασική αρχή, δηλαδή ο έλεγχος της συμβατότητας ενός νόμου, είτε είναι αυτός ενός κανόνα, είτε είναι νόμος, είτε είναι ε, διοικητική πράξη, είτε είναι συνταγματικός κανόνας. Για το διοικητικό για το νομοθετικό κανόνα, για το νόμο δηλαδή, ο δικαστής δεν μπορεί να εφαρμόσει και καλείται να μην εφαρμόσει νόμο ο οποίος αντίκειται σε διεθνή διάταξη ιεραρχικά ανώτερη και αυτό έχει οριστεί από το ανώτατο αναιρετικό δικαστήριο του Βελγίου για πρώτη φορά στην Ευρώπη με την περίφημη απόφαση της 27ης Μαΐου του 1971 Λουσκή ε, και είναι πρώτη φορά που απαγγέλλεται η ιεραρχική υπεροχή του διεθνούς κανόνα και η άμεση εφαρμογή του στο, στην εσωτερική ενωμή τάξη. Τα δικαστήρια λοιπόν δεν θα αναγνωρίσουν ουδεμία συνέπεια και εφαρμογή νόμου που θα επιβάλλει μέτρα ασφαλείας ασύμβατα κρινόμενα φέρυπιν, φέρυπιν με διάταξη τη σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών. Όταν νόμος παραβιάζει θεμελιώδες δικαίωμα το, οποίο εγγυάται ταυτόχρονα δε το σύνταγμα μια χώρα και διεθνή σύμβαση όπως η Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τουλάχιστον όσον αφορά το Βέλγιο, το συνταγματικό δικαστήριο το ίδιο παρεμβαίνει για να ακυρώσει τον νόμο αυτόν ή για να τον κηρύξει αντισυνταγματικό στο πλαίσιο ενός προδικαστικού ερωτήματος απόφαση της 11ης Ιουνίου του 2015 και κύριε Πρόεδρε, εάν ξεπεράσω το χρόνο μου, μην διστάσετε να μου σηκώσετε ένα κόκκινο πανί. 11 λοιπόν Ιουνίου του 2015, απόφαση του Σταγματικού Δικαστηρίου του Βελγίου, που δίνει ένα παράδειγμα προστασίας των θεμελιωδών ελευθεριών και αναφέρομαι σε απόφαση του Σταγματικού Δικαστηρίου του Βελγίου, η οποία απόφαση αποτελεί τη συνέχεια της αποφάσεως της 8ης Απριλίου του 2014 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της Digital Rights Ireland Limited του 2014, Απρίλιο 2014. Πρόκειται για απόφαση αρχής και πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα. Σε αυτήν την απόφαση αρχής λοιπόν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου ακυρώνει οδηγία. Την οδηγία της 15ης Μαρτίου του 2006, τη λεγόμενη οδηγία περί διαφυλάξεως δεδομένων οδηγία η οποία υποχρέωνε τον παρέχοντα υπηρεσία τηλεπικοινωνίας ε, ηλεκτρονικής, διαδικτύου και τα λοιπά, πρόσβαση δηλαδή για το κίνημα του διαδικτύου, ήταν υποχρεωμένο όσο παρέχουν αυτήν την υπηρεσία να διαφυλάσει μία σειρά δεδομένων που παρήγαγε ο χρήστης του. Γιατί ήταν απαραίτητο αυτό για να παραμένουν οι ε, πληροφορίες αυτές στην διάθεση και για χρήση αστυνομικών ερευνών για την καταπολέμηση τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Το δικαστήριο του Λουξεμβούργου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου, έκρινε πως η υποχρέωση για διακράτηση των δεδομένων αυτών για ορισμένο χρονικό διάστημα δεδομένων σχετικών με το προσωπικό βίο των ιδιωτών σορευόμενη με τη δυνατότητα πρόσβασης των αρχών στη βάση αυτών δεδομένων συνιστούσε βαρύ, βαρία παρέμβαση στο δικαίωμα για την προστασία του ιδιωτικού βίου, στο δικαίωμα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπω τα περιγράφουν τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Πρόκειται για μια βαρία παρέμβαση, λέει λοιπόν το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Και ταυτόχρονα αυτή η βαρία παρέμβαση ελέγχει και την αναλογικότητα, μάλλον το δικαστήριο ελέγχει την αναλογικότητα της παρέμβασης αυτής και μας λέει ότι δεν είναι αναλογική αυτή η παρέμβαση γιατί και εδώ ορίζει κάποια στοιχεία. Μιλάει δηλαδή για το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, γιατί ήταν υπερβολικά ευρύ, γιατί αναφέρεται σε άτομα ακόμα για τα οποία δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι μπορεί να έχουν αναπτύξει τρομοκρατικές ή εγκληματικές δραστηριότητες, γιατί επίσης δεν υπάρχει καμία εξαίρεση για τον ε, δεσμευόμενο από το επαγγελματικό απόρριτο γιατί δεν υπάρχει καμία υλική ή δικονομική εγγύηση για την προστασία των δικαιωμάτων των διδών. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν ακυρώνεται οδηγία και να τελειώνω εδώ πρόεδρε. Δύο λεπτά ακόμη. Πολύ ωραία και αυτή, η απόφαση, λοιπόν, αυτή την απόφαση έρχεται το, το δικαστήριο του, το σταγματικό δικαστήριο να την εφαρμόσει ουσιαστικά ακυρώνοντας τον βελγικό νόμο μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της εν λόγω οδηγίας. Αυτό αποτελεί παράδειγμα εφαρμογής του κράτους δικαίου. Και ολοκληρώνω βέβαια, δεν ελέγχονται μόνο οι νομοθετικές πράξεις αλλά και οι διοικητικές, όπως και το ίδιο το Σύνταγμα το ίδιο το Σύνταγμα κρίνεται, γιατί στο Βέλγιο έχουμε κρίνει και κρίνουμε ότι το ίδιο το Σύνταγμα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις θεμελιώδεις αρχές και ελευθερίες που εγγυώνται οι διεθνείς συμβάσεις. Το ίδιο το Σύνταγμα πρέπει να σύμμορφούται στις εγγυήσεις που έχουν, ε, στα δικαιώματα που εγγυώνται οι διεθνείς συμβάσεις και αν το κρίνετε απαραίτητο μπορώ να σας προσφέρω και σχετικά παραδείγματα. Πρόεδρε ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας και κλείνω με μία μόνη φράση. Η δικαιοσύνη δεν είναι εξουσία του κράτους. Η δικαιοσύνη είναι εξουσία της δημοκρατίας. Πιστεύω, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Uh, Δυστυχώς ήμασταν πολύ απλόχεροι όσον αφορά το χρόνο που δώσαμε στους πρώτους ομιλητές, οπότε η επόμενη θα πρέπει να είναι σύντομη. Ο Μίκλος Σάντο έχει τώρα το λόγο, είναι διαχειριστικός διευθυντής και επικεφαλής του Τμήματος Αναλύσεων του Κέντρου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, μέλη των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, κυρίες και κύριοι, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και να τα πω απλά. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Είμαι ευγνώμων προς όλους τους ευρωβουλευτές και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές που οργάνωσαν την ακρόαση για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα που είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Είμαι νομικός Ούγκρος και υπεύθυνος του Ινστιτούτου για τις αναλύσεις που γίνονται όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε στη σύντομη παρουσίασή μου θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στους κινδύνους που ελοχεύουν από ένα θεσμοθετημένο μηχανισμό κράτους δικαίου. Όταν μιλάμε για μια τέτοια διαδικασία που τυποποιεί, που θεσμοθετεί το μηχανισμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, βρίσκω τρεις παράγοντες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν οποιοδήποτε τέτοιο τέτοιο μηχανισμό υποχρεωτικό θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πρώτα απ' όλα η ίδια η σύλληψη του, των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων και υπάρχει και θέμα νομιμότητας. Τέτοια προβλήματα είναι πολύ πιθανόν να εμφανιστούν άπαξ και θεσμοθετηθεί ένας τέτοιος μηχανισμός. Θέλω εδώ επίσης να υπογραμμίσω ότι τέτοια προβλήματα δεν θα προκύψουν ε, μόνο όσον αφορά τα όργανα που θεσπίζουν την νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη, αλλά και στο δικαστικό σώμα όσον αφορά την ε, συμμόρφωση, της δικαστικές αποφάσεις και την εφαρμογή τους. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, δύο λόγια για την ε, ασάφεια της έννοιας του κράτους δικαίου. Ακριβώς επειδή υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις, επειδή δεν υπάρχουν οι ίδιες ιστορικές εμπειρίες, δεν υπάρχει σαφής και συγκεκριμένος παγκόσμιος ούτε καν ευρωπαϊκός ορισμός για το τι είναι. Η επικοινομορφία των προσεγγίσεων έχει να κάνει επίσης και με τις διαφορετικές γλώσσες, οι οποίες διατυπώνουν την εξουσία αυτή. Κράτος δικαίου, Ρέχστατ... Ε, rule of law κλπ. Διατυπώνεται διαφορετικά δηλαδή στις διάφορες γλώσσες. Και έχει και ιδεολογική σημειολογία διαφορετική. Τι θα μπορούσε να σημαίνει. Σημαίνει οτιδήποτε τα δικαστήρια ή άλλα όργανα συμμόρφωσης στο νόμο θέλουν να σημαίνει. Είναι μια έννοια η οποία εξελίσσεται συνεχώς εδώ λοιπόν θα ήθελα να παραθέσω κάτι που αναφέρεται σε ένα από τα έγγραφα εργασία της Μπάρμπαρα Σπινέλη, Ευρωβουλευτού, που αναφέρει κάτι που λέει η Επιτροπή της Βενετίας και λέει ότι υπάρχουν δυσκολίες προκειμένου να εφαρμοστεί το κράτος δικαίου σαν μια ανεξάρτητη και ουσιαστική έννοια. Και μάλιστα φαίνεται να πρόκειται για κάποιες υποθέσεις πολύ περισσότερο από ότι για μια σαφώς ε, αρχή η οποία εφαρμόζεται με σαφήνεια και συγκεκριμένα. Όντως υπάρχει κάποια ευελιξία εδώ και αυτό φαίνεται και πάρα πολύ καλά από την ε, πρακτική του σταγματικού δικαστηρίου έτσι όπως ε, τροποποιήθηκε. Οι νομοθέτες, το κοινοβούλιο, το rule of law το κράτος δικαίου το θεωρούν σε μια αφηρημένη έννοια που έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά του κράτους. Το συνταγματικό δικαστήριο λοιπόν το ερμήνευσε σαν μια προδιαγραφή που εφαρμόζεται κατά περίπτωση. Συνεπώς το δικαστήριο διασφαλίζει ότι κρατάει τον τζόκερ, ότι δηλαδή μπορεί να δράσει σαν συνημοθέτης τελικά. πως αυτή η ασαφής έννοια μπορεί τελικά να χρησιμοποιηθεί σαν πολιτικό εργαλείο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανένας δεν ξέρει τι ακριβώς σημαίνει, πώς να μετρήσει το κράτος δικαίου. Μπορεί κανείς να το μετρήσει. Αν προσπαθήσει, είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιηθούν μηχανισμοί οι οποίοι τελικά θα οδηγήσουν σε πολιτικές πιέσεις ή σε κριτική στην πολιτική η οποία εφαρμόζεται. Και αυτό φαίνεται και από τις δράσεις της Επιτροπής και επιπλέον αυθαίρετη εφαρμογή μιας τέτοιας διαδικασίας θα μπορούσε να οδηγήσει στην παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας από τα ευρωπαϊκά όργανα γιατί θα αφαιρούσε συνταγματικές ε, αρμοδιότητες από τα κράτη-μέλη που δεν έχουν ε, παραχωρήσει ακόμα τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς να αποπολιτικοποιήσουμε και την ε, προσέγγιση αυτή. Γιατί τελικά όντως αφαιρούνται εξουσίες από τα κράτη-μέλη και υπάρχει κίνδυνος πολιτικοποίησης. Το θέμα της κυριαρχίας πάντως θα οδηγήσει σε συγκρούσεις δικαιοδοσίας ανάμεσα στα δικαιοδοτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκείνα των χωρών μελών. Υπάρχουν διαφορετικά συνταγματικά δικαστήρια και για χρόνια τώρα υπάρχει το επιχείρημα του τελικά ποιος είναι πιο κατάλληλος να ερμηνεύσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία και σε τι βαθμό. Το είδαμε αυτό και στη Γερμανία με δικαστικές αποφάσεις εκεί ή με άλλες που συνεχίζονται ακόμα όσον αφορά ποσοστώσεις που βρίσκονται στο Ουγγρικό, για παράδειγμα, συνταγματικό δικαστήριο. Θα καταλήξουμε σε καυγάδες για την νομιμότητα επίσης. Υπερεθνικά όργανα μη αιρετά θα αμφισβητήσουν την νομιμότητα πράξεων που θα έχουν αποφασιστεί από αιρετά όργανα. Ένας τέτοιος λοιπόν μηχανισμός χωρίς να υπάρξει αλλαγή στις συνθήκες δεν είναι μια καλή ιδέα. Είναι κάτι που θα αμφισβητηθεί κατά πολύ στο εγγυσμένο. δεν θα υπάρχει η βάση της νομικής διαδικασίας που να διαθέτει νομιμότητα. Έπειτα υπάρχει το θέμα της υπευθυνότητα και της ευθύνη. Πώς εφαρμόζεται το κράτος δικαίου στα κράτη-μέλη. Υπάρχει η δυνατότητα παραβιάσεων, αλλά τα σώματα ε, συμμόρφωση στο νόμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρουμε αν θα είναι εκείνα ή εκείνα των κρατών μελών που θα μπορούν να επιβλέψουν αποφάσεις και διαδικασίες που έχουν να κάνουν με το μηχανισμό αυτό τον ευρωπαϊκό Κράτος δικαίου. Είναι πάντα θέμα ερμηνείας. Ποιος αναλαμβάνει αυτή την ερμηνεία. Θα πρόκειται για ένα διακυβερνητικό όργανο που θα αποτελείται από τις χώρες μέλη, οπότε οι χώρες μέλη με αυτόν τον τρόπο επανακτούν κυριαρχία. Μια τέτοια διαδικασία θα δημιουργούσε όλο και περισσότερα ερωτήματα. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας θα μπορούν να παρέμβουν στην αναπομείνουσα κυριαρχία των χωρών μελών και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα τη αντιμετώπιζαν εξωτερικές ε, πιέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Και αν υπάρχει χρόνος, ευχαρίστως να απαντήσω στις ερωτήσεις και στα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα τον ε, λόγο στον τελευταίο ομιλητή, είναι ο κύριος Νταρίου Ζαβιστόφσκι ο οποίος ε, προέρχεται από το Εθνικό Συμβούλιο της Δικαιοσύνης στην Πολωνία και είναι και μέλος του Ευρωπαϊκού ε, Δικτύου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ε, εκτιμώ την πρόσκληση που μας έχετε αποστείλει έτσι ώστε το Εθνικό Συμβούλιο Δικαιοσύνης στην Πολωνία να συμμετάσχει στην συζήτηση. Ε, εμείς ε, θα, εγώ στην διάρκεια της ε, παρέμβασής μου θα αναφερθώ στον τρόπο με τον οποίο το Εθνικό Συμβούλιο Δικαιοσύνης της Πολωνίας προσπίζεται την ανεξαρτησία του καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται με τον ενωσιακό νόμο κυρίως δε ε, όσον αφορά το άρθρο 6 ε, της ε, συνθήκης και το άρθρο 46 και το άρθρο 47 συγγνώμη, της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Εμείς θεωρούμε ότι η προστασία του ατόμου είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό θα σας δώσω δύο παραδείγματα. Ε, προστασία της, του δικαιώματος της ιδιοκτησίας ε, που αναφέρεται άλλοτε, άλλωστε και στο άρθρο 17 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι κομμουνιστικές αρχές κρατικοποίησαν, εθνικοποίησαν όλες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ε, ε, μέχρι 50 εκτάρια. Αυτό ήταν ε, μια κατάφορη παραβίαση των δικαιωμάτων τους και βεβαίως είχαν την δυνατότητα αυτοί οι άνθρωποι να ζητήσουν αποζημίωση, πράγμα το οποίο κατάφεραν να κάνουν μετά το 1999, γιατί μέχρι τότε δεν είχαν καμία δυνατότητα να ε, επιζητήσουν ε, τέτοια ε, αποζημίωση. Θεωρήθηκε δηλαδή τότε force majeure και δεν ακολούθησε καμία δικαστική διαδικασία για την αποζημίωση. Επίσης, ένα δεύτερο παράδειγμα, η ευθύνη της ε, ε, διοίκησης ε, για ενδεχόμενη ζημία που έχει λάβει η χώρα τα δικαστήρια είναι ε, ανεξάρτητα ε, και επομένως ε, χρησιμοποίησαν την νομοθεσία με αναδρομική ισχύ για το θέμα αυτό. Αυτά είναι δύο καλά παραδείγματα τα οποία δείχνουν ότι στην Πολωνία ε, μετά την αλλαγή του 1999 ε, είχαμε την δυνατότητα να ε, εισάγουμε την αρχή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης στο Σύνταγμα. Ε, ο διαχωρισμός ε, των ε, τριών εξουσιών αναφέρθηκε σαφώς στο Σύνταγμα και επίσης δημιουργήθηκε και το Εθνικό Δικαστήριο της Δικαιοσύνης στην Πολωνία ακριβώς έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της ε, της δικαιοσύνης. Έχει δε μεταξύ των καθηκόντων του ε, και την αρμοδιότητα ορισμού των ε, δικαστών. Αυτό θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι δίνει πλήρες εξουσίες στο, στις δικαστικές αρχές. Ωστόσο, εάν διαβάσει κανείς προσεκτικά την, το, Σύνταγμα ε, τότε θα καταλάβει ότι και η νομοθετική και η εκτελεστική εξουσία έχουν την δυνατότητα να επηρεάσουν ε, την ε, δικαστική. Μετά την μεταπολίτευση είχαμε 20 υπουργούς δικαιοσύνης και ο καθένας από αυτούς ήθελε να μεταρρυθμίσει το δικαστικό σύστημα αλλά ε, είχαμε και έναν ε, ε, Υπουργό Δικαιοσύνη ο οποίος έκλεισε 79 από τις πρωτοβάθμιες δομές μετά την παρέτησή του ξαναδημιουργήθηκαν αυτές οι δομές, ανακλήθηκαν λοιπόν οι αποφάσεις του. Ναι, υπάρχει και το, το συνταγματικό δικαστήριο ε, ε, ε, στα πλαίσια του οποίου έχει έχει υπάρξει εμπλοκή ε, λόγω της, ε, του ορισμού των ε, μελών του, του δικαστηρίου αυτού. Έχει υπάρξει τροποποίηση του, του τρόπου λειτουργίας και του τρόπου διορισμού των δικαστών και αυτές οι αλλαγές αντιτίθενται στο άρθρο 2 του συντάγματος έχουν ε, υπάρξει πολλές ε, ε, κινήσεις για τον έλεγχο της συνταγματικότητας των αποφάσεων αυτών καθώς επίσης ε, και της ανεξαρτησίας ε, του ε, δικαστηρίου. Πρέπει να σας πω ότι έτσι όπως έχουν τα πράγματα και αν δεν υπάρξει κάποια αρχή, συγγνώμη, αν δεν υπάρξει κάποια συνταγματική διασφάλιση, τότε ενδεχομένως στο μέλλον θα αντιμετωπίσουμε περιπτώσεις όπου το δικαστήριο θα παραλύσει. Πολλές είναι οι δυνατές λύσεις. Το σημαντικό πάντως ε, είναι ε, να υπάρχει συνταγματικός έλεγχος απέναντι στις ε, αποφάσεις της νομοθετικής ή εκτελεστικής εξουσίας. Είναι σημαντικό να ακούει η εξουσία την φωνή του κόσμου και θα πρέπει ε, να είναι υπόλογοι ε, απέναντι ε, στη, στα μάτια του κόσμου. Θα πρέπει οι πολίτες να καταλαβαίνουν ότι και να έχουν πλήρη διασφάλιση ότι η νομοθετική εξουσία και η εκτελεστική εξουσία δεν μπερδεύεται με την δικαστική στην πράξη συχνά συμβαίνει πολιτικοί ή οι άνθρωποι των μέσων ενημέρωσης να σχολιάζουν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης θεωρώντας ότι αυτό είναι ένα προνόμιο των δικαστών. Αλλά αυτό είναι προζημίαν των δικαστηρίων. Επομένως, ε, θα πρέπει να εξηγηθεί στον κόσμο ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης ε, είναι ε, πολύ σημαντική για την διασφάλιση δίκαιης δίκης και οπωσδήποτε ε, θα πρέπει να ε, προχωρήσουν οι αρχές αυτές ε, με τις άλλες διασφαλίσεις και εχέγγυα που παρέχονται από την δικαιοσύνη. Θα ήθελα να υπογραμμίσω εδώ ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης μπορεί να έχει και πρακτικές συνέπειες. Αυτό ε, συζητήθηκε ε, στην, ε, στα πλαίσια της σύμβασης της Βενετίας καθώς επίσης και στα πλαίσια της δικαστικής συνεργασίας αλλά εξακολουθεί να είναι λίγο μακρινό θέμα για, του, για τον απλό κόσμο. Η γνωμοδοτήσεις μπορεί να μην είναι σαφές ε, και μπορεί να αναφέρονται σε διαφορετικά στοιχεία της ανεξαρτησίας μπορεί να αναφέρονται ε, στον ορισμό των δικαστών, μπορεί να αναφέρονται στα οικονομικά, μπορεί ε, να αναφέρονται σε πολλά στοιχεία. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι να καταλάβουμε τι είναι σημαντικό για τον κόσμο όταν αναφέρονται στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης βλέποντας ε, τις αποφάσεις ε, του ε, Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέποντας τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Στρασβούργου, καθίσταται σαφές ότι θα πρέπει να διασφαλιστούν τα ελάχιστα κοινά πρότυπα επί των οποίων να βασιστεί και ο δικαστής για να κάνει σωστά τη δουλειά του γιατί μπορεί να υπάρχουν διαφορές ε, στα δικαϊκά συστήματα των διαφόρων χωρών, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές. Ε, όσον αφορά τώρα τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα μπορούσε κανεί να σκεφτεί ότι θα ακουστεί περισσότερο η θέση του, του ε, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου από ότι επιμέρους δικαστηρίων. Ε, γι' αυτό λοιπόν και κατά αυτή την έννοια ίσως θα ήταν καλό ε, να κυκλοφορήσουν και από πλευράς του Κοινοβουλίου ε, κάποια ελάχιστα πρότυπα, στο έγγραφο δηλαδή του Κοινοβουλίου να συμπεριληφθούν και αυτά τα κάποια ελάχιστα πρότυπα τα οποία μπορούν να καλύψουν τον ε, έλεγχο ε, ε, της, τον έλεγχο που μπορεί να έχει η νομοθετική και η εκτελεστική εξουσία επί της δικαστικής. Και βεβαίως ένα μεγάλο κεφάλαιο είναι η εφαρμογή των προϋποθέσεων και των προτύπων. Θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει ε, και τις ετήσιες εκθέσεις ε, που προετοιμάζουν τα κράτη-μέλη ε, για να περιγράψουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η δικαστική εξουσία. Αυτό θα μπορούσε να ενισχυθεί και να διευρυνθεί. Θα ολοκληρώσω κυρία Πρόεδρε λέγοντας το εξής. θέλω να υπογραμμίσω ότι εμείς έχουμε γραπτό υλικό το οποίο θα μπορούσε να σας φανεί χρήσιμο. γιατί εμείς σαν Εθνικό Συμβούλιο έχουμε πολλές γνωμοδοτήσεις προς το Συνταγματικό Δικαστήριο της Πολωνίας που ίσως ε, σας, ε, είναι, σας φανούν χρήσιμες. Επίσης, νομίζω ότι ε, μαζί και με τους άλλους δικαστές ε, θα μπορέσουμε να σας, ε, απο, να σας ε, απαντήσουμε στα ερωτήματά σας. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Τώρα, ερωτήσεις. Και μετά θα ακούσουμε τις απαντήσεις. Η Σόφιν Χετφάλτ είναι η πρώτη που έχει ερώτηση. Ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα προς τον κύριο Μπόμπεκ. Είπατε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε ήδη στη διάθεσή μα. Συμφωνώ απόλυτα και αυτό είναι και ο στόχο της έκθεσή μου. Να μην επανεφεύρουμε τον τροχό, αλλά πρέπει να εντοπίσουμε και κενά, αδυναμίες. Αναφερθήκατε στις διαδικασίες ε, επί κυρώση, επί παραβάση, συμφωνώ μαζί σα, αλλά δεν νομίζω ότι τέτοιες διαδικασίες επιβαραβάσει έτσι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα καλύπτουν και όλα τα ζητήματα. Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Γιατί εσείς αναφέρατε παραδείγματα σε συγκεκριμένη χώρα μέλος, με την πάυση δικαστών και το άλλο είχε να κάνει με την ελευθερία του τύπου. Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν ακριβώς ότι κάτι λείπει, ότι υπάρχει ένα κενό γιατί το εργαλείο που χρησιμοποιείται είτε είναι αυτό των οπτικουστικών, η οδηγία δηλαδή, είτε εκείνη για την απασχόληση, δεν διασφαλίζουν απόλυτα την ανεξαρτησία ε, του δικαστικού ή την ελευθερία του τύπου. Είπατε επίσης άρθρο 2 θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν ε, φτάνει για τη διαδικασία παραβάσης. Αυτό θα ήθελα να επεκταθείτε περισσότερο παρακαλώ. Δεύτερη ερώτηση. Είπα και στην αρχή ποια είναι η κατάσταση στις Ηνωμένε Πολιτείε με τον ορισμό του νέου δικαστή στο Supreme Court, στο Νότο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτείων, που έχει πολιτικοποιηθεί πολύ. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, γιατί δεν υπάρχει ευρωπαϊκή κυβέρνηση που ορίζει τους δικαστές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' αυτά, επρόκειτο για 28 νέους δικαστές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Ήμουνα υπέρ του να αυξηθεί το νούμερο, αλλά το ότι πρόκειται για 28 δείχνει ότι οι κυβερνήσεις θεωρούν ότι έχουν τον δικό τους δικαστή, παρόλο που οι δικαστές θα έπρεπε να είναι εντελώς ανεξάρτητοι. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κανείς να μην σκεφτεί ότι υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στον αριθμό των δικαστών και το πώς τους βλέπουν τα κράτη-μέλη. Αλλιώς δεν θα ήταν 28 αυτοί οι δικαστές απαραίτητα. Τώρα, και για σας και στον κύριο Τεκότ θέλω να ρωτήσω κάτι. Και να απαντήσω λιγάκι και στα σχόλια του κύριου Ζαβιστόφσκι. Τι κάνετε εάν, για παράδειγμα, η δικαστική εξουσία ή το κράτος μέλος δεν είναι αντικειμενικό. Τι μέσα υπάρχουν για να παρεύουμε. Ο κύριος Τεκότ είπε το Σύνταγμα, οι νόμοι δεν μπορεί να αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο. Ναι, αλλά δυστυχώς αυτό συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις. Οπότε τι κάνουμε τότε. Και προς τον κύριο Σάντο, κοιτάξτε, μια γενική παρατήρηση μόνο μπορώ να κάνω. Εσείς δεν δέχεστε το γεγονός ότι υπάρχουν οι συνθήκε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι υπάρχουν συμφωνίες όπου υπερισχύει το ευρωπαϊκό δίκαιο του εθνικού δικαίου και όχι μόνο στις περιπτώσεις που αναφέρατε. Το δέχεστε αν πρόκειται για παράνομες κρατικές επιχορηγήσεις ή για παραβίαση περιβαλλοντικών ε, νόμων. Αλλά όχι πάντα φυσικά έχετε δικαίωμα να έχετε ό,τι άποψη θέλετε, αλλά αν δεν δέχεστε κάποια κυριαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε πρόβλημα. Τέλος, είπατε ότι είναι ασαφής η έννοια του κράτους δικαίου. Σε ένα βαθμό ίσως, αλλά όχι ότι δεν έχει και νόημα. Και ακούσαμε την δικαστή Νισμπέργκερ που είπε ότι έχει νόημα. Ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε κοινά στοιχεία ώστε από την ομολογία να προχωρήσουμε στον ορισμό του κράτους δικαίου. Αλλά όλη η ιδέα του να έχουμε ένα μηχανισμό που να περιλαμβάνει όχι μόνο κυρώσει, αλλά προηγουμένω διάλογο για το πώ θα αποφεύγουμε καταστάσει που θα οδηγήσουν σε κυρώσει, θα μπορούσε να περιλαμβάνει ένα κοινό ορισμό, την εκπόνηση ενό κοινού ορισμού όσον αφορά το κράτο δικαίου. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Παύλο Ράτζι. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα και εγώ να ρωτήσω κάποια πράγματα. Ε, δεν ξέρω αν θα απαντήσουν οι καλεσμένοι μας, θα το αποφασίσουν εκείνοι αυτό. Λοιπόν, κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι το πλαίσιο του δικαστικού συστήματος μιας χώρας είναι ένα πράγμα και άλλο πράγμα είναι το πώς λειτουργεί αυτό. Αυτά δηλαδή είναι δύο ζητήματα που οδηγούν σε αυτό ακριβώ το δίλημα, ότι δεν είναι το ίδιο. Στη χώρα μου, για παράδειγμα, το δικαστικό σύστημα είναι αρκετά καλό. Όμως, αργεί τόσο πολύ στην λειτουργία του, προκειμένου να ανταποκριθεί στους πολίτες, να χρησιμοποιήσει τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους οι πολίτες, καταλήγει τελικά στο να μην λειτουργεί. Κατά κάποιο τρόπο τουλάχιστον. Οπότε ναι, ανεξαρτησία του συστήματος, ποιότητα δικαστών βεβαίως. Αλλά δυστυχώς αποφασίζει με τεράστια καθυστέρηση. Και είναι εντελώ διαφορετικό να αποφασίσει το δικαστικό σύστημα και να βρίσκει λύσει σε μία διένεξη μετά από 4-5 χρόνια και άλλο να καταλήγει αμέσω. Έπειτα, αυτά που είπε ο κύριο Ντεκότ για την οικονομική ηλική ανεξαρτησία. είναι πράγματι πολύ σημαντικό κατά κάποιο τρόπο να αντιγράψουν οι ευρωπαϊκές χώρες αυτό που ισχύει στο Αμερικανικό Σύνταγμα, ότι δηλαδή το οικονομικό καθεστώς των δικαστών είναι κάτι που εγγυάται το σύστημα ανεξαρτήτως πολιτικών αποφάσεων. Υπάρχει δηλαδή μια ρήτρα διασφάλισης. Πολύ σημαντικό αυτό. Το είδα όταν είχαμε την Τρόικα στην Πορτογαλία, όπου έγιναν περικοπές σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και οι δικαστές δεν είναι στην πραγματικότητα δημόσιοι υπάλληλοι, γιατί ναι μεν ανήκουν σε ένα συνταγματικό σύστημα, παρόλα αυτά πλήγησαν και δικοί τους οι μισθοί. Η κυβέρνηση δηλαδή ήθελε να περιορίσει και τη δικιά τους ε, οικονομική κατάσταση. Αυτό όμως πρέπει να το προστατεύσουμε. Υπάρχει όμως κάτι διαφορετικό, όπου δεν συμφωνώ με τον κύριο Ντεκότ. Και αυτό είναι η λογιστική κατάσταση. Εγώ δεν νομίζω ότι το δικαστικό σύστημα πρέπει να διαθέτει όλα τα μέσα για να έχει ένα δικό του διοικητικό σύστημα, αυτό θα ήταν επικίνδυνο. Γιατί τότε θα βρισκόμασταν σε μια άλλη αρνητική κατάσταση. Θα ήταν ένα άλλο ελάττωμα της δημοκρατίας, γιατί θα είχαμε φτιάξει την κυβέρνηση της δικαστικής αρχής, των δικαστών. Επικίνδυνο για τη δημοκρατία αυτό. Και ιδιαίτερα για τη δικιά μας δημοκρατία, τις δικές μας δημοκρατίες. Γιατί τώρα έτσι όπως έχουν τα νομικά μας συστήματα είναι τόσο περίπλοκα όπου οι δικαστές έχουν τεράστια εξουσία διότι ερμηνεύουν ένα ιδιαίτερα περίπλοκο νομικό σύστημα. Άρα η ελευθερία τους όχι μόνο να καταλήξουν όσον αφορά τα γεγονότα αλλά να προχωρήσουν και στην εξέβρεση λύσεων του προσφέρει μια τεράστια εξουσία, πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχουν κατά το παρελθόν. Και έτσι έρχομαι στο τρίτο μου ζήτημα. Κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Πώς θα δώσουμε δημοκρατική νομιμότητα στη δικαστική εξουσία. Εγώ πιστεύω ότι ιδιαίτερα σε ένα σύστημα όπως είναι το ευρωπαϊκό νομοθετικό σύστημα, όπου είναι ένα σύστημα και ισλό, όχι βάση του ρωμαϊκού δηλαδή δικαίου. Η δυνατότητα αποφάσεων και αποφάσεις των δικαστών έχουν μεγαλύτερη ισχύ. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει ένας τρόπος για να οδηγηθούμε σε δημοκρατική νομιμότητα. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να αντιγράψουμε το αμερικανικό σύστημα. Ούτε λέω ότι πρέπει να είναι αιρετοί οι δικαστές. Όμως, κατά πάσα πιθανότητα θα έπρεπε στην περίπτωση των δικαστών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου, για παράδειγμα λέω, να υπάρχει ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ψηφίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μια ψηφοφορία προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία. Γιατί ακόμα και στην περίπτωση των χωρών δεν είναι τόσο ένα θέμα κομμάτων, είναι ένα θέμα... Είναι ένα θέμα σύλληψης του κόσμου, νοτροπίας. Αυτό λοιπόν με φέρνει στην τελευταία μου παρατήρηση. Προς τον κύριο Τσάντο. Με εκπλήσει η ιδέα αυτή ότι το κράτος δικαίου είναι κάτι ασαφές. Διότι η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, η παράδοση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που είναι στη βάση του κράτους δικαίου, δεν είναι τίποτα το ασαφές. Αν κάποιος από την Ουγγαρία από τον Αντρέτο δεύτερο της Ουγγαρίας έχουμε κάτι σαν μάγνα κάρτα που μιλά για το κράτος δικαίου και υπάρχει. Οπότε το κράτος δικαίου είναι μια τεράστια έννοια, πολύ σημαντική, που όταν κανείς έχει να αποφασίσει για θεμελιώδη ζητήματα, ζητήματα μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιήσει το κράτος δικαίου. Έχουμε διάφορες μάγνα κάρτα ανά τον κόσμο. Είτε πρόκειται για τη Γαλλία ε, του 1789, είτε πρόκειται για άλλα και στην Ουγγαρία και αλλού. Υπάρχει τέτοια παράδοση των Ευρωπαίων ήδη εδώ και πάρα πολύ καιρό και στην Ουγγαρία. Οπότε μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό που είπατε. Πρόεδρος. Σύντομο παρακαλώ. Ναι, θα είμαι σύντομος. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πολύ τους ε, ομιλητές μας. Για τον Βέλγο δικαστή, θέλω να το ρωτήσω στην ερμηνεία που κάνει της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος. Δέχεται ότι μπορεί να ορίσει από το κοινοβούλιο το σώμα των δικαστών, ότι δηλαδή η εξουσία η δικαστική να υποβάλλεται στην ε, λαϊκή ετοιμιγορία. Δέχεται δηλαδή ότι μπορεί να είναι συμβατό κάτι τέτοιο με την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος εάν οι δικαστές του ε, δικαστικού σώματος στον νότο του δικαστηρίου εκλέγονται από το Κοινοβούλιο, από την εκτελεστική εξουσία. Και κάτι τώρα να ρωτήσω τον κύριο Πόροκο όσον αφορά την, επικαιρότητα για κάτι που αποφάσισε το δικαστήριο τη εβδομάδα αυτή. Η Χάρτα Θεμελιδών Δικαιωμάτων μπορεί να πληγεί από συμφωνίες όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και όσον αφορά τα, την ισότητα κοινωνικών δικαιωμάτων για τους Ευρωπαίους εργαζόμενους το Ηνωμένο Βασίλειο μετά τη συμφωνία αυτή που έχουμε τώρα. Μπορεί να αλλάξουν οι προδιαγραφές με την συμφωνία αυτή που έγινε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να ξέρουμε κατά πόσο παραβιάζεται η Χάρτα Θεμελιδών Δικαιωμάτων από τη συμφωνία ακριβώς αυτή με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστούμε κυρία Ρεβόλαλον. Ευχαριστώ και πολύ σύντομα. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα του σεβασμού του κράτους δικαίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί και εγώ ε, ξαφνιάστηκα όταν άκουσα πως θεωρείται ότι το κράτος δικαίου είναι ασαφές και έχει επαρκώς προσδιορισμένο. Βέβαια αυτό συμφωνεί και με την ιδέα ότι δεν είναι δυνατόν απλώς να εφαρμοστεί το κράτος δικαίου διότι αυτή τη στιγμή μηχανισμοί του, η δικαιοδοτική για το σεβασμό του κράτους δικαίου είναι δυσκίνητη και δυσεφάρμοστη. Είναι κάτι το οποίο προκύπτει λοιπόν και φέτος, όταν μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις σε ορισμένα ζητήματα και βέβαια ακούω κάποιες ιδέες ότι ίσως να ήταν σκόπιμο να δίνονται πεστροκίνητρα παρά κυρώσεις. Ωστόσο από άλλες διατάξεις εξίσου σημαντικέ με τις αξίες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρομαι σε ζητήματα οικονομικά, βρίσκουμε τον τρόπο να εφαρμόσουμε μια σειρά μηχανισμών, το Συμφώνο Σταθερότητας και εκεί λειτουργούν οι κυρώσεις και κάποια κράτη μάλιστα εκλήθησαν να τις αντιμετωπίσουν. Ο λόγος λοιπόν για τον οποίο υποστηρίζω απολύτως τις θέσεις της ε, ε, συναδέλφου Νετφέλτ είναι αυτό ότι πρέπει να δοθεί κανονιστικό κανονιστικός χαρακτήρας στο κράτος δικαίου ώστε κανείς πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην μπορεί να σκεφτεί ότι οι αρχές και οι αξίες μας είναι ασαφείς η πρόεδρο Μας έχουν μείνει τέσσερα λεπτά για τον κάθε ένα από τους ομιλητές μας. Ας ξεκινήσουμε ανάποδα. Εσείς παρακαλώ, κύριε Ζαβιτόφσκι, για τέσσερα λεπτά μόνο. Ναι, πολύ σύντομα θα προσπαθήσω να τοποθετηθώ τα θέματα της ε, ευθύνης και υπευθύνοντας της δικαιοσύνης ένα ζήτημα το οποίο προκύπτει και θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτή η αρχή σημαίνει πως έχει την ευθύνη ο δικαστής για τα όσα πράττει. Αυτό ισχύει στο πολωνικό δίκαιο. Εάν φερθεί ανεύθυνα δηλαδή, προκύπτει ευθύνη του και αναλαμβάνει δράση το πειθαρχικό συμβούλιο με βάση αρχές του πειθαρχικού δικαίου. Εάν παραβιάσει αρχές της διοντολογίας ένας δικαστής, συμπεριφερθεί κατά τρόπο παράνομο, μπορεί να ε, υποστεί και, και ποινικές κυρώσεις. Όλα αυτά είναι εγγύησεις που εξασφαλίζουν με την απέτηση ο, το Πειθαρχικό Συμβούλιο να είναι σύμφωνο με το ποινικό ε, δικαστήριο την ανεξαρτησία του δικαστή. Και μάλιστα υπάρχει και δυνατότητα προσφυγής προς αποζημίωση όταν έχουν εκδοθεί ε, ορισμένου τύπου αποφάσεις. Όταν δηλαδή δεν είναι σύμφωνες ε, οι δικαστικές αποφάσεις με τις αρχές του δικαίου μπορεί να πάει ο διάδικο σε ένα αστικό δικαστήριο για να ζητήσει αποσημείωση για μια κακή δικαστική απόφαση. Δεν μπορεί λοιπόν να ισχυριστεί κανείς ότι δεν θα έχει ευθύνη ο δικαστής για τα όσα πράττει. Θέλω να το πω αυτό είναι σημαντικό και θα το τονίσω. Πρέπει να γνωρίζει κανείς πώς έχει λάβει μια απόφαση ο δικαστής και πώς διορίζεται ως δικαστής. Η Διεθνής Ένωση Δικαστών τόνισε εδώ πως η η επιλογή αυτή πρέπει καταρχάς ε, να, να ανήκει, καταρχήν να ανήκει στη δικαιοσύνη. Ωστόσο πρέπει ορισμένα ζητήματα να λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή των προσώπων που θα απαρτήσουν το δικαστικό σώμα και ιδιαίτερα για τον πρόεδρο ο οποίος ορίζει τις ε, θέσεις τις οποίες θα καταλάβουν οι δικαστές και θα πρέπει και όπως είπαμε ορίζει τον δικαστή στην κάθε θέση. Αυτά είναι τα σημαντικότερα ζητήματα που προκύπτουν από το Εθνικό Δίκαιο. Ο κύριος Σαντρό, πρόεδρε ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς θα χρειαστεί να φύγω μόλις ολοκληρώσω τα σχόλιά μου γιατί έχω ένα αεροπλάνο για τις 8.30. Εν συντομία. Μάλλον εγώ φταίω, αλλά φαντάζομαι με παρερμηνεύσατε γιατί εγώ μιλούσα για τον ορισμό του κράτους δικαίου. Βεβαίως και γνωρίζω το κράτος δικαίου έχει διάφορες, διάφορα συνιστώσεις και διάφορα στοιχεία. Καλύτερα συνισταμένες και στοιχεία. Ωστόσο, κωδικοποιημένη έννοια ή καλύτερα ορισμός του κράτους δικαίου χρειάζεται. Αυτό είναι βασική αρχή του δικαίου, είναι πολύ ευέλικτο και γι' αυτό αναφέρθηκα και στην ε, ε, νομολογία του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ουγγαρίας ε, που έχει προσπαθήσει να ενθαρρύνει και να ενισχύσει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου ακόμα και εις βάρος της ελευθερίας της έκφρασης σε μια περίπτωση όταν όμως θεώρησε ότι είναι πιο σημαντική η ελευθερία της έκφρασης, τότε προήγαγε την ελευθερία της έκφρασης εις βάρος ε, της αξιοπρέπειας του ανθρώπου και αυτό είναι ένα ζήτημα ευελιξίας του ορισμού του κράτους δικαίου όπως ήθελα να εξηγήσω και όπως θα μπορούσαν να ερμηνεύουν τα δικαστήρια ανα πάσα στιγμή. Και χωρίς ορισμό δεν μπορεί να προσμετρηθεί η έννοια του κράτους δικαίου ή το καθεστώς του κράτους δικαίου. Και έτσι θα υπάρχει κίνδυνος κοινωνικής μηχανικής και Παρέμβαση κάτι το οποίο μετά το κομμουνιστικό, μετά το κομμουνιστικό καθεστώς δεν χρειάζεται η Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Ζοντεκότς. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Έχω σημειώσει αρκετέ ερωτήσει. Θα προσπαθήσω πάρα πολύ σύντομα, μια και έχω στεθεί μου λίγα λεπτά μόνο, για την κυρία Νετφέλτ που μας ρωτάει τι πράττουμε σε περίπτωση που δικαιοδοτική αρχή κράτους μέλους πάβει να είναι αντικειμενική και τι εννοείται κυρία Ιντφέλτ με το αντικειμενική γιατί στην πραγματικότητα εάν η απόφαση της δικαιοσύνης δεν είναι νόμιμη, ε, ακυρώνεται. Αν η απόφαση του δικαστή ενός δικαστή είναι μεροληπτική, αν ίσως αυτό εννοείται ως μια αντικειμενική, τότε θα ε, κληθεί στην τάξη, θα ανακληθεί στην τάξη ο δικαστής ή θα, θα εξωτερωθούν οι συνέπειες της αποφασής του. Υπάρχει ένα σύστημα, ένας μηχανισμός προσφυγών Ίσως δεν απαντώ όμως αυτό που ρωτάτε. Κύριε Νετφέλτ. Ναι, αλλά μας είπατε ότι ο νόμος, το Σύνταγμα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διεθνείς διατάξεις, με τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου. Ε, τι κάνουμε λοιπόν, γιατί εγώ βλέπω πολλές περιπτώσεις νόμων της εθνικής νομοθεσίας αντίθετες κατάφορα με τη διεθνή ε, νομοθεσία και πολλές φορές και συντάγματα φαντάζομαι μπορεί να περιέχουν ρήτρε αντίθετε με το διεθνέ δίκαιο, χωρί μικρόφωνο ο δικαστή. Λοιπόν, στην ε, εσωτερική ένωμη τάξη δεν θα δοθεί η παραμικρή συνέπεια, δεν θα αναγνωριστεί η παραμικρή συνέπεια στην αντίθετη με τη διεθνή τάξη ένωμη διάταξη. Ε, παραδείγματι, η προσωρινή κράταση στο εσωτερικό βελγικό δίκαιο είναι 24, 24 ώρε ανά το όριο. Υπάρχει το άρθρο 5 της Σύμβασης των Δικαιωμάτων. Στο βελγικό δίκαιο προτείνεται σε περίπτωση τρομοκρατικών ε, ε, αδικημάτων, σχετικών με τρομοκρατία αδικημάτων, να παραταθεί αυτό. Υπάρχει η πρόταση να παραταθεί το όριο της προσωρινής κράτησης ε, μέχρι και στις 72 ώρες. Τώρα αν αυτό πάει αντίθετα με σχέση στην Διεθνή Συνθήκη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη μάγνη Κάρτα που λεγόταν νωρίτερα, θα αρνηθεί να εφαρμόσει το σχετικό, το σχετικό νόμο ο δικαστής στη Γαλλία, το Συμβούλιο Επικρατείας, το Γαλλικό, το Conseil ΤΑ συγκεκριμένα και το Συνταγματικό Συμβούλιο, τα αυτά όργανα έχουν ακυρώσει μέτρα κατοίκων περιορισμού ή προσωρινής, ε, προσωρινού κλεισίματος ε, ε, καταστημάτων για λόγους ισλαμιστικής προπαγάνδας, η συμμετοχή σε τρομοκρατικές ισλαμιστικές δραστηριότητες, γιατί τα καταγγελόμενα περιστατικά δεν ε, υποτάσσονταν σε αρχές αντικειμενικότητα και τι προδιαγραφέ του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάτι αντίστοιχο με το κράτο δικαίου υπάρχει στη Γαλλία. Για δεν συμφωνώ καθόλου με τον κύριο Σαντόρο. Υπάρχει κράτο δικαίου. Είναι ξεκάθαρο, δεν έχω αρκετό χρόνο για να το εξηγήσω. Υπάρχει κράτος δικαίου και λειτουργεί στις χώρε μα και είναι αναγνωρίσιμο με βάση αυτές τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας Γαλλίας και του Συνταγματικού της ε, Συμβουλίου. Η κύρωση λοιπόν για την ασυμβατότητα είναι η άρνηση από τον Εθνικό Δικαστή να δώσει έννομες συνέπειες. Είναι τεράστια αυτή η εξουσία και υπάρχει. Ο υπήκος, ο διάδικος ο οποίος ε, επικαλείται αυτή το ασυμβίβαστο έχει την προστασία του ε, ιστορικού δικαστή. Κύριε Ραντζέλ, και εσείς διατυπώσατε μια αντίστοιχη ερώτηση. Λέγατε ότι η βραδιποροί δικαιοσύνη στο εσωτερικό σύστημα δεν προχωρούν εγκαίρως ε, οι δικαστικές αποφάσεις. Βεβαίως, πρώτη αδικία είναι αυτό, να κρατάει υπερβολικά μακρό διάστημα μια δίκη. Πέραν αυτού έχουμε την εγγύηση του ευλόγου, ε, της ευλόγου διάρκειας και συστηματικά καταδικάζονται οι χώρες μας σε περίπτωση καθυστέρησης υπερβολικής στην απόδοση της δικαιοσύνης, αλλά έχω να σας ξαναστείλω και το μπαλάκι, να σας επιστρέψω το μπαλάκι, γιατί υπάρχει δυνατότητα να οργανωθεί το δικαστικό σύστημα, ώστε να μην κατακλείονται από ανοησίες οι δικαστικές αρχές. θεριπίν, μπορεί να φτάσει στη χώρα σας μία ε, παράβαση για ε, παράνομη στάθμευση μέχρι το ανώτατο συνταγματικό, το δικαστήριο. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν τρόποι να οργανωθεί η δυνατότητα προσφυγή στη δικαιοσύνη ώστε να μην έχουμε τέτοιε υπερβολικέ και καταχρηστικέ προσφυγέ. Επίση, για το υλικό καθεστώ των δικαστών θα συμφωνήσω μαζί σα στι παρατηρήσει και εξάλλου έχουμε καταθέσει το Συμβούλιο της Ευρώπης τις παρατηρήσεις μας για ό,τι θεωρούμε πως αποτελεί παραβίαση της αρχής αυτής της ηλικής ανεξαρτησίας. Τώρα ίσως να μην καταλάβατε πολύ καλά γιατί είπατε ότι δεν συμφωνείτε μαζί μου και παραθέτω τα λόγια σας. Δεν θεωρώ πως η δικαστική εξουσία πρέπει να έχει την αυτοδιοικητική ανεξαρτησία για, την, για τα επιμελητιακά. Μα προφανώς θα συμφωνήσουμε κύριε ε, βουλευτά. Η βελγική κυβέρνηση όμως θέλει κάτι τέτοιο και βεβαίως και έχετε δίκιο όταν λέτε ότι μπορεί αυτό να αποτελεί απειλή. Επίσης με ρώτησαν ε, εάν έχω κάποια αντίρρηση στο να αποφασίζει ο λαός ως προς τους διορισμούς των δικαστών και αν οι διορισμοί των δικαστών θα μπορούσαν να αναπόκειται στο δικαστήριο αν έχω αντίρρηση γι' αυτό. Αγαπητοί πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, δεν πρόκειται να φτύσω μέσα στη σούπα που με έθρεψε. Εγώ εξελέγην ως πρόεδρος στην θέση αυτή τη δικαστική που έχω από την γερουσία τη Βελγική. Άρα προφανώς και θεωρώ ότι θα πρέπει ένα κοινοβούλιο να έχει λόγο στον διορισμό. Βέβαια όσον αφορά το δικό μου προσωπικά το διορισμό δεν υφίστανται πλέον αυτές οι διατάξεις και το σύστημα ανήκει πια στην ιστορία για το Βέλγιο αλλά υπάρχουν ένομε τάξεις όπου ένα το συμβούλιο δικαστικό ε, απαρτίζεται όχι μόνο από δικαστές. Στο Βέλγιο έχουμε δικαστές κατά το ίμιση στο Συμβούλιο αυτό, πολύ ενδιαφέρον, να μπορεί και ο δικαστής να τοποθετείται για τους υποψηφίους και κατά το ίμιση από μέλη της κοινωνίας των πολιτών που ορίζει το, ε, η γερουσία. Άρα βεβαίως ε, μπορεί άμεσα ή έμεσα ένα κοινοβουλευτικό όργανο να ε, τοποθετείται όσον αφορά τον διορισμό των δικαστών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, στην αρχή θεώρησα ότι θα έχω μόνο δύο λεπτά, αλλά βλέπω ότι... Ε, λοιπόν, το άρθρο το οποίο αναφέρατε δεν καλύπτουν τα πάντα. Ναι, βεβαίως, συμφωνώ με αυτό που λέτε. Ωστόσο, μπορώ να απαντήσω διτά. Πρώτον, όπως ήδη αναφέρθηκε από την κυρία Νιουσμπέργκερ, οι δικαστές είναι στη θέση τους για να ε, βρίσκουν λύση ε, σε υποθέσεις. Εγώ είμαι πεπερασμένος, όχι όσον αφορά το πνεύμα μου, αλλά όσον αφορά τη θέση που έχω. Δεν μπορώ να λύσω τα πάντα τα οποία δυνάμει θα μπορούσα να λύσω από αυτή την άποψη. Γι' αυτό ζητώ να βλέπουμε συγκεκριμένε υποθέσεις, γιατί σε αυτές τις, ε, μέσω αυτών των συγκεκριμένων υποθέσεων μπορώ εγώ να δω εάν και κατά πόσον έχει υπάρξει ε, παραβίαση δικαίου. Δεύτερο, πέρα από το συνταγματικό ε, ε, νόμο, δηλαδή ακούστηκε ή υπονοήθηκε από πολλούς το ζήτημα είναι να δούμε εάν έχουν υπάρξει συστημικές παραβιάσεις ε, του, νόμου ή του δικαίου στις ε, χώρες. Ε, Μία τέτοια απόφαση όμως η οποία θα ελαμβάνεται κεντρικά πιστεύω ότι θα ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ας πούμε σκεφτείτε την... την την απόφαση Ζολάγκε ε, και πόσο μπορούσε κανείς ε, διτά να την ε, ερμηνεύσει. Και το σημαντικό, το είναι να δούμε πώς θα μπορούσε να είχε αποδειχθεί. Είναι ευρύτερο λοιπόν το πρόβλημα. Δεύτερη ερώτηση, άρθρο 2 της χάρτας να σας πω, σε αυτή την περίπτωση εγώ αναφέρθηκα στο έγγραφο εργασίας 5 και την γνωμοδότηση της κυρίας Σπινέλη, η οποία λέει η ίδια ότι το άρθρο 2 φαίνεται να μην ε, είναι αρμόδιο από αυτή την άποψη. Πάντα θα πρέπει να κινούμαστε ε, στο πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου. Το άρθρο 2, ε, όπως και το άρθρο 51 της ε, χάρτας, ε, λένε, αναφέρουν ότι θα πρέπει να υπάρξει και δευτερογενές δίκαιο βάσει το οποίο να οδηγηθεί ένα θέμα, μια υπόθεση μάλλον στο δικαστήριο. Αλλά δεν έχουν συστατική ερμηνεία όλοι αυτοί οι νόμοι. Αυτή είναι η πρώτη απάντηση. Η δεύτερη απάντηση το άρθρο 2, όπως και η χάρτα, είναι σημαντικά όταν έχει περάσει κανείς ε, το, βήμα, το πρώτο βήμα. Όταν θα έχω βρει τη βάση, τότε βεβαίως ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι ώστε να καθορίσω πόσο σημαντική είναι η παραβίαση κτλ. Δηλαδή θα πρέπει πρώτα να έχει τη νομική βάση και μετά να περάσει την πόρτα. Μέχρι να περάσει την πόρτα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ε, η μεταρρύθμιση του πρωτοδικείου ε, νέες δικαστικές διαδικασίες ε, ε, σχετικά με τη διεύρυνση του πρωτοδικίου, όχι του δικαστηρίου, είναι σωστό να πει κανείς ότι οι διαδικασίες είναι διαφορετικές και και να πω εδώ ε, παρεπιπτόντως ότι το δικαστήριο έχει πολύ ε, ε, ευεργητηθεί από τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου για τις οποίες τον το ευχαριστούμε. Τώρα όσον αφορά το τι κάνουμε όσον αφορά την πραγματική την πραγματική λογοδοσία, ε, τότε κανείς μπορεί να κάνει τις δικές του επιλογές. Είδαμε και το, το παράδειγμα το οποίο αναφέρατε προηγουμένως των ΗΠΑ. Τελευταίο ε, ερώτηση έχει φύγει ο ενδιαφερόμενος, αλλά νομίζω ότι ο κύριος ε, Τόντο επίσης το υπέβαλε. Ε, ίσως δεν τα διάβασα όλα, ε, και δεν έχω διαβάσει ε, πολύ συγκεκριμένα τα στοιχεία της ε, πρόσφατης συμφωνίας και επομένως και της απόφασης του Συμβουλίου και δεν πρόλαβα να διαβεστώ. Επίσης όταν αναφέρθηκα σε έλεγχο προδικαστικών ερωτημάτων στο δικαστήριο πρέπει να σας πω ότι αυτά είναι δύσκολα ε, τα, ε, οι αποφάσεις αυτές ε, θα πρέπει να έρχονται εκ των υστέρων με την έννοια ότι θα πρέπει τα εθνικά δικαστήρια να έχουν ήδη μια πρώτη αξιολόγηση επί της οποίας θα γνωμοδοτήσει το δικαστήριο. Από αυτή την άποψη έχω υπάρχει ένα πρόβλημα, ε, είναι δύσκολο με τους υφιστάμενους κανόνες να φτάσει στο δικαστήριο ε, αυτό το θέμα. Αυτά θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ε, διερμηνείς, να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στην στην ακρόαση αυτή και να ζητήσω από τους ε, Πολωνούς ε, δικαστές εάν ε, έχουν κάποιο υλικό το οποίο ανέφεραν στην παρέμβασή τους να μας το αφήσουν. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που ήρθατε και που είσαστε μαζί μας.